Sí. Καθίστε παρακαλώ, λέει πρόεδρο. Καλημέρα προ όλου. Καλά, καλησπέρα. Αρχίζει επομένω η συνεδρίαση τη Επιτροπή Αγγλία. Και πρώτα-πρώτα θα πρέπει να εγκρίνουμε τη μέση διάταξη. Επίση θα πρέπει πρώτα-πρώτα να σα πω ότι έχει γίνει κάποια ελαφρά αλλαγή στη μέση διάταξη. Το θέμα το οποίο αφορά την πειρατεία στον Ινδικό δεν θα ζητηθεί σήμερα όπως προβλεπόταν ε, διότι όπως μας εξηγήθηκε η Επιτροπή Άμυνας Ασφαλής και Μεταφορών και η δική μας πρόκειται να κάνουν από κοινού μια συνεδρία για να συζητήσουν αυτό το θέμα στις 16 Ενδεκάτου. Οπότε και θα έρθει και ο αντινάβαρχος Πίτερ Χάτσον. Οπότε θα έχουμε έτσι οι δύο υποπιτροπέ και η επιτροπή ε, μια κοινή ζήτηση όσον αφορά την πειρατεία στον ειδικό. Οπότε, στη θέση αυτού του θέματο πρόκειται να συζητήσουμε την παρουσίαση της τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό που αφορά το Γενικό Συμβούλιο Αλληλείας στη Μεσόγειο. Ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον δυνατό να ζητηθεί αυτό το θέμα, αντί για εκείνο το θέμα τη μεσδιάταξη θα γίνει, επαναλαμβάνει πρόεδρο η συζήτηση για το Συμβούλιο της ε, Αιλία. Σε επίσης πρέπει να σα βυσμάνω ότι η σημερινή συνεδρίαση ε, μεταδίδεται παντού, ούρμπι ετόρμπι, μέσω της Τωσέλωσης Κοινοβουλίου. Τώρα, θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων τη 20ης και 21 η του Ιουλίου. Και αν το τέλο συνεδρίαση ουδή έχει κάτι, να προτείνει ως ένσταση, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται πρακτικά. Κατά τρίτον, έχουμε τις ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Σας ανακοινώνω ότι έχουμε διαβάσει με email όλους με ένα κατάλογο, μια, μια αλληλογραφία εκ μέρους της γραμματείας της Επιτροπής μας και στο Εδιμβούργο πρόκειται να γίνει μια διάσκεψη όπου θα υπάρχουν εκπρόσωποι των ΡΑΚ για να συζητήσουμε τι θα γίνει με την μεταρρύθμιση στον κλάδο της αλληλείας και της κοινής ελευθερικής πολιτικής το 2012. Ζητήσαμε από τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Στίβενσον, να μας εκπροσωπήσει, άλλωστε είναι Σκοτσέζος που μα εκπροσωπήσει στη διάσκεψη του Εδιμβούργου. Επίση, πρέπει να σα ενημερώσω ότι την επόμενη Δευτέρα στι 5 Δεκάτου θα γίνει συνεδρίαση Ιντερ Rax. Εδώ στι Βρυξέλλε. Και με την αδειά σα θα προσκαλέσω εαυτήν στη διάσκεψη. Αυτό προσκεφτώ λοιπόν για να πάω εκεί πέρα και έτσι για πρώτη φορά, ας πούμε για πρώτη φορά, θα παραστώ όχι ως βουλευτή αλλά ως πρώτη φορά ω πρόεδρο σε αυτή τη ε, διάσκεψη του τεράξει, επαναλαμβάνει πρόεδρο. Επίση, κατά τέταρτον, στην ημερησία διάταξη έχουμε την ψήφιση τη Συμφωνία Ελληνική. Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Διορθώνει το γραμματέα. Πρώτο πρώτο, ναι, ναι το Έχουμε την αλληλευτική σύμπραξη τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Δημοκρατία τη Γουινέα. Κάτι το οποίο προβλέπεται να ψηφιστεί σήμερα. Επίσης, όπως ήδη έχει συζητηθεί για μακρόν, θα πρέπει να δώσω το λόγο στον συνάδελφο που ζήτησε να μιλήσει. Tack så väldigt mycket. Eh, saker och ting har förändrats i Guinea vi har diskuterat den här frågan. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη φορά συζητήσαμε το θέμα Έγινε πραξικόπημα στη Γουινέα όμως. Εν μεταξύ. Περιμένω να βάλει τα ακουστικά της κυρία Φράγκα. Όπως ξέρετε, έγινε πραξικόπημα έλεγα στη Γουινέα. 23 Δεκεμβρίου πέρσι έγινε. Και τώρα έχουμε μια κυβέρνηση που δεν είναι δημοκρατική. Και το καθεστώς με τον κύριο Μοζακαμπάρα, το συνταγματάρχη Μοζακαμπάρα, έσφαξε τουλάχιστον 150 άτομα στο Κονακρί. Σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Χιλιάδες ε, τραυματίστηκαν. Συστηματικοί βιασμοί έγιναν και θέλουμε να μπορέσουμε να συζητήσουμε την αλληλευτική συμφωνία πριν ψηφίσουμε. Διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα, είναι θέμα αρχής. Η Γαλλία σχεδιάζει να αποσύρει τη βοήθεια που χορηγεί προς την χώρα αυτή και θα ήταν παράξενο η Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δοθήσεις της παρούσεις καταστάσεις να υπερψηφίσει τη συμφωνία όταν δεν γνωρίζουμε σε τι θα εξυπηρετήσει η υπηρεσία μας. Ή μάλλον ξέρουμε σε τι θα, θα, εξυπηρετήσουν τα χρήματά μας. Θα τροφοδοτήσουν ένα καθεστώς που βασανίζει τον πληθυσμό. Θα πρέπει να, ψηφίσουμε, να το συζητήσουμε και ψηφίσουμε. Um, äh, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε συνάδελφος. Όντως ε, πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι συμβαίνει τελικά στη Γουινέα και κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα, μπορούμε να περιμένουμε αύριο έτσι ώστε να το κάνουμε στην επόμενη συνεδρίαση, να μας πληροφορήσει δηλαδή και κάποιος από την Κομισιόν να μας πει τι γίνεται στη Γουινέα. Φυσικά μέχρι την τελευταία τελική ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια θα πρέπει να έχουμε συζητήσει, να έχουμε καταλήξει σε μια α, θέση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Στίβενσον έχει το λόγο. Πρόεδρε, συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπαν οι συναδελφοί και συμμερίζομαι το ότι η Γουινέα δεν είναι και το υπόδειγμα δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, έχουν ε, αποθέματα αλλιευτικά τα οποία μπορούν να θέσουν σε εμπορία. Αν εμεί πληρώνουμε για, αυτές, για τα αποθέματα, για αυτούς τους πόρους, εφαρμόζουμε με τον πιο αυστηρό τρόπο την αλλιευτική συμφωνία που έχουμε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι που στέλνουμε καταλήγουν στην διατήρηση των αποθεμάτων, στο να ε, μπορούν να αλλιεύουν οι ντόπιοι ψάρια και να τρέφονται να εξασφαλίσουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αλλιεύματα για επεξεργασία. Αν σταματήσουμε αυτή τη συμφωνία για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και αν είναι απολύτως θεμητός, θα, όλοι αυτοί οι πόροι οι αλληλευτικοί θα καταλήξουν στα χέρια των Ρώσων ή των Κορεατών που θα έρθουν και δεν θα ενδιαφέρονται καθόλου για την απασχόληση των ντόπιων, για την διατήρηση των αποθεμάτων, δεν θα ενδιαφέρονται καθόλου για όσα ενδιαφερόμαστε εμείς. Θα υπάρξει υπεραλίευση και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν ψάρια. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ψαρέψουν τα πάντα μέχρι να μην υπάρχει ούτε ένα ψαράκι στη θάλασσα. Εμείς μπορούμε με τις ελληνικέ συμφωνίες μας να ελέγξουμε τα πράγματα και να εργαστούμε με έναν πολύ επαγγελματικό τρόπο. Οπότε μην νομίζετε ότι κάνοντας αυτή την πολιτική χειρονομία εδώ στην Επιτροπή μας, ψηφίζοντας δηλαδή κατά τη συνέχεια της συμφωνίας θα λύσουμε το πρόβλημα έλλειψης δημοκρατίας στην Γουινέα ούτε θα λύσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα που νομίζουμε ότι μπορούμε να, λύσουν, να λύσουμε. Έχουν πόρους ελευτικούς, θα βρουν κάποιον άλλο να τους πουλήσουν. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Δημιουργεί ακόμη χειρότερες καταστάσεις για τους ε, αλληλείς που ζουν στις ε, απομακρυσμένες παράκτιες περιοχές. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν ε, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι θίγουμε το θέμα αυτό, αλλά ε, συμφωνώ με ακούστηκαν, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι επιπλοκές, γιατί νομίζω, Πρόεδρε, ότι ε, Έχουμε αυστηρό χρονικό χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό λάβατε την απόφαση να, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αν εμεί καθυστερήσουμε, τι επιπτώσει θα έχει η Επιτροπή Αλίας, ας το σημειώσουμε ας πούμε σήμερα, ότι αποφάσισε να περιμένει ε, για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι έγινε στην ε, Γουινέα. Πρέπει βεβαίως κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα να λάβουμε μια απόφαση, ξέροντας όμως και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχει επιφυλάξει η Επιτροπή Ανάπτυξη. Αυτό έχω να σα πω. Όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Και υπογραμμίσαμε την πρόθεση τη ε, Επιτροπή, τι ανησυχίε μα μάλλον, για τη διαφθορά στη Γουινέα και την έλλειψη νομιμότητα του καθεστώτο. Σαν απλή Ήρθα για να πω ότι υπάρχει πρόβλημα συνοχής όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ασυνέπεια μεταξύ αναπτυξιακής πολιτικής και των άλλων εξωτερικών. Και δεν μπορεί να περάσει μια λευτική συμφωνία με πληρωμή 300.000 ευρώ σε, μια, ε, σε ένα καθεστώς που βιάζει τις γυναίκες και σκοτώνει. Διότι αυτά τα χρήματα θα τους χρησιμεύσουν να αγοράσουν ξυφολόγχες. Θα ήθελα να υποστηρίξω εκ βάθους καρδίας με μεγάλη αποφασιστικότητα τις προτάσεις που έκανε η προλαλήσασα και οι προλαλήσασες. Δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό μήνυμα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια ήπειρο ειρήνη και συμφιλιώσεω και συνεργασία, την επομένη μιας τέτοια μεγάλη φαγής, να είναι μια ψήφο συνεργασία. που θα την συνάψουμε κλείνοντας τα μάτια απέναντι σε μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πλέον στοιχειωδών. Ε, Κύριε Στίβενσον, λυπούμε, αλλά δεν είμαστε εμείς που θα επιβάλλουμε τη δημοκρατία στη Γουινέα, αλλά το να δεχθούμε και με κλειστά τα μάτια μια αλλιευτική συμφωνία την επομένω του δράματος δεν μπορεί παρά να τις πιο αντιδημοκρατικές και βίες μεθόδους. Η Ευρώπη πρέπει να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα την επομένη όταν το, θύμα, τον θυμά, το αίμα των θυμάτων ακόμα χνίζει. Κυρία Αντινόρο. Κύριος Αντινόρο. Κυρία Πρόεδρε, Καταλαβαίνω τους λόγους και καταλαβαίνω συνάδελφοι τους λόγους για τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε τα τραγικά γεγονότα. Πιστεύω όμως ότι η πολιτική πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες ε, πρέπει ε, να λαμβάνει υπόψη αυτά τα σημαντικά, να δεν πρέπει να υπερισχύει τόσο σημαντικών ζητημάτων. Εκ μέρου ΕΛΚ πρέπει να πω, δεν μπορώ να πω θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε. Δεν θα σε εκπλήσει ότι θα ζητούσα να αναβληθεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί η ψηφοφορία, διότι αργότερα σαν ομάδα να συνεννοηθούμε, διότι δεν μπόρεσα να συνομιλήσω με τους άλλους συναδέλφους. Μόλις φτάσαμε στις Βρυξέλλες όλοι σήμερα. Να έχουμε κάποιο χρόνο να συναντηθούμε τα μέλη της ομάδας, ήταν κάτι χρήσιμο για να συζητήσουμε το θέμα. Καταλαβαίνω ότι μέχρι αύριο δεν θα έχουμε νέες πληροφορίες τα ίδια σήμερα όπως και αύριο θα είναι. Δεν θα έχουμε άλλες πληροφορίες. Δεδομένου ότι στη Γουινέα έγιναν αυτά που έγιναν. Έχουμε δικτατορία στη Γουινέα. Θέλω να επιθυμίσω στον συνάδελφο Στίβενσον κάτι. Να παραμείνει η συμφωνία είναι να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια χρήματα που δεν έπρεπε να τους δώσουμε σε αυτό το καθεστώς επειδή επικρατεί σύγχυση και δεν έχω ξεκάθαρε ιδέε ούτε εγώ τι συνάδελφοι, να αναβάλουμε για το πρωί για να ξεκαθαρίσουμε τι ιδέε και να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε το θέμα με του συναδέλφου. Μετά το τέλο τη Επιτροπή και να αποφασίσουμε απόψε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο το πρωί. Δεν ζητώ να μην ψηφίσουμε τη συμφωνία. Απλώ ζητώ μια μικρή αναβολή για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και ξεκαθαρίσουμε τι ιδέε. Για να ξέρουμε ξεκάθαρα τι κάνουμε. Sí, eh, ε, por parte Μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρίσταται η κυρία Σαβαρή, η οποία και έχει το λόγο. Oui, merci, la... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι. Να ξεκινήσω από τον τελευταίο αγορητή. Αύριο υπάρχει ευκαιρία να μπορέσετε εις λεπτομέρεια να τα δείτε όσον αφορά τις αληφτικές συμφωνίες. Οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει η ενημέρωση αυτή, μια που σήμερα το πρωί τα είπαμε στην πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνση Ανάπτυξης οι οποίοι παρέστησαν στη συνέντευξη αυτή και καταλήξαμε ότι θέλουμε να σας πούμε ότι παρακολουθούμε από κοντά τι εξελίξει και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε το πώς εξής τα πράγματα, όπω κάνετε και εσείς όσον αφορά τα θέματα τα πιο τεχνοκρατικά σε σχέση με την διαδικασία αυτή. Ναι, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, αναβολή της ψηφοφορίας. Ε, ίσως το θέμα φτάσει μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο το Συμβούλιο θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει τελικά να εγκρίνει τον λόγο κανονισμό. Ούτω ώστε να μπορέσουμε να για την οικονομική αντιστάθμιση. Που θα είναι 1 εκατομμύριο 50.000 ευρώ. Οπότε και έτσι θα υπάρξει η, η φόρους στήριξη του κλάδου. Δύο φορές. Ε, έχουν ζητηθεί οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής. Οπότε, καθ' τον τρόπο, αν εδώ βάλετε κατά δύο μέρες ε, την ψήφιση, θα, καταρθίσουν και οι εκταμιεύσεις κατά δύο μέρες, οι 25, ε, όπως ξέρετε τώρα, παρακολουθούν αποθαλάσσεις το τι γίνεται στην Γουινέα, γιατί οι διπλωμάτες δεν βρίσκονται στην πόλη, δεν μπορούν λόγω του κινδύνου. Και η γενική μας διεύθυνση, επομένω δεν έχει περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια. Και τα πράγματα εξελίσσονται. Οπότε και αυτές οι πληρωμές, οι καταβολές, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να γίνουν. Είτε έχουμε αναβολή, είτε όχι. Είτε έχουμε διακοπή, είτε όχι. Γιατί έχουμε άλλωστε και κάποιου είδου προθεσμίε για, τη, για τη σχετική κοινοποίηση, ειδοποίηση, όχληση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τι μείζονε αλλαγέ τολισμό, όσον αφορά την πολιτική που θα ασκηθεί και άρα για το κατά πόσον θα συναυθεί αυτή η ε, συμφωνία και να δούμε μετά πού θα βαδίσει η κοινή αλληλευτική πολιτική. Επίσης, έχουμε και κάποια ανάλυση από πλευράς δημοσιονομικής, από πλευράς ε, νομικής, ε, γιατί υπάρχει εδώ πέρα και μια πολιτική διάσταση που δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Μια που η Κομισιόν και ίσως θέλουν να, να συμπληρώσουν και οι συνάδελφοι Γενικής Διεθνή ε, Ανάπτυξης για να μας πούν τι γίνεται όσον αφορά ε, τις εξελίξεις σε σχέση με το άρθρο 96 και έχουμε ε, μετά από 48 ώρες από αυτή τη σφαγή τα πράγματα φυσικά και είναι πάρα πολύ λεπτά και δύσκολα. Οπότε έχει δημοσιεύσει λοιπόν ότι τόσο χρόνο μα μένει αν θέλει να κάνει την αναβολή εφορία, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση των συνέπειών. Μια που βεβαίω όλοι οι εμπλεκόμενοι αλλά και το Κοινοβούλιο πρόκειται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αυτή τη αναλύσεω. αυτό μπορώ να σα πω, αλλά είμαι στη διάθεσή σα. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, gibt es also... εάν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αναβολή για τον Νοέμβριο. Θα ήθελα να το ζητήσουμε αυτό και θα πρέπει να λάβουμε και από την Κομισιόν αλλά και από άλλα βήματα πληροφορίες για το τι σημαίνει αυτό. Ίσως αν μπορούσαμε αύριο να έχουμε τις πρώτες πληροφορίες να μπορούμε να δώσουμε και ένα μήνυμα μη υπογράφοντας αυτή την ε, ε, συμφωνία. Πρέπει να αναλύσουμε λοιπόν όλα τα δεδομένα και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πάμε τον Νοέμβρη και να έχουμε έτσι τον απαραίτητο χρόνο ως τότε για να μπορέσουμε να πληροφορηθούμε επαρκώς για το τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Señora Lobán. Eh, Ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα πρέπει να λάβουμε και άλλες πληροφορίες όσον αφορά την αληφτική συμφωνία με τη Γουινέα. Διάβασα την αξιολόγηση που αφορούσε την τελευταία συμφωνία με την Γουινέα. Διάβασα, σας λέω, την ανάλυση την ανεξάρτητη ανάλυση που διενεργήθηκε από σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας συστήνω να διαβάσετε το κείμενο. Στο κείμενο αναφέρεται σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανένα έλεγχο όσον αφορά την χρήση των χρημάτων. Μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε σε, αυτό, σε αυτή τη σύμβαση, παραδείγματος χάρη την υποστήριξη των μικρών αληφτικών εκμεταλλεύσεων μπορούμε να έχουμε μακρύ κατάλογο σημείων που δεν γίνονται σεβαστά. Αυτό έγινε στο παρελθόν, ενώ είχαν αναλυφθεί κάποιες υποχρεώσεις. Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι γίνονται αυτά τα χρήματα. Δοθήσεις της παρούσης καταστάσεως, δοθέντος του καθεστώτος, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει αυτό καθόλου. Πρόκειται περί που έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, λιγότερο από ένα χρόνο, και όλος ο κόσμος έκανε σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ποιες είναι οι συνέπειες όλων αυτών. Έχουμε ένα εκατομμύριο ευρώ, αυτό συζητούμε, και δεν θέλουμε να φτάσουν στα χρήματα ενός δικτάτορα. Εδώ μας είπατε για κάποιο αλληλευτικό που ψάρευε στα νυχτά της Γουινέας, που δεν είναι δεδειγμένη στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που συμβαίνουν στην ξηρά. Αν διαβάσετε τις εφημερίδες, θα δείτε ότι γίνονται πολλές σφαγές. Φτάνει να δείτε τι έγινε στο ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Κονακρί. Όλους αυτούς τους βιασμούς, τα βασανιστήρια, κατά αθώων. Δεν μπορούμε καθόλου να ψηφίσουμε αυτό το σημείο σήμερα. Πρόεδρος. Γκάλερ. President, I certainly would not approve taking decision. Πρόεδρε, ας μην λάβουμε απόφαση σήμερα. Θα ήθελα να ξέρω ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους απλούς ανθρώπους. Για τα σκάφη επίσης που θέλουν να μας διαθέσουν ίσως αφορά ανθρώπους και ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Μπορεί να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, Μπορεί να το κάνουμε μετά από σήμερα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για κάτι. Εγώ δεν έχω συμφέροντα όσον αφορά τα σκάφη, δεν ξέρω τι σκάφη υπάρχουν εκεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε. Να ξέρουμε όμως μέχρι αύριο το πρωί ποιες είναι οι συνέπειες. Μας είπαν ότι πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα, λόγω του κατεπήγοντος του θέματος. Μπορούμε να φύγουμε όμως από εδώ να, εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτά που συμβαίνουν στη Γουινέα, αλλά τελικά αν εμείς δεν υποστηρίξουμε τη συμφωνία θα την πληρώσουν ίσως άλλοι και όχι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις φρικαλαιότητες. Κύριε Στίβενς, συμφωνώ με τον κύριο Γκάλαρ. Όσο άσχημο και δυσάστο αυτό είναι το καθεστώς, δεν έχει σημασία. Θα βρουν τα χρήματα για να πουλήσουν τους αλευτικού πόρους. Θα καταστραφούν όμως οι αλευτικοί πόροι. Οι Ρώσοι, οι Κορεάτες θα καταφτάσουν, θα τους δώσουν ένα εκατομμύριο ευρώ για τα ψάρια και τα αλευτικά δικαιώματα, θα καταστρέψουν τα αλευτικά αποθέματα και οι απλοί άνθρωποι που ήδη υποφέρουν κάτω από αυτό το καθεστώς το βίο καθεστώς θα δουν ότι δεν τους έχει μείνει ψάρι, λέπει να ψαρέψουν. Εν τω μεταξύ θα έχουμε κάνει μια πολιτική χειρονομία, θα έχουμε αρνηθεί αλληλευτικά δικαιώματα σε 25 από τα δικά μα αλευτικά σκάφη και θα βοηθήσουμε να καταστραφεί και ο ελευτικός τομέας της Γουινέα για τους απλούς ανθρώπους, τους απλού ψαράδε, τι αλευτικέ κοινότητε που ζουν στι ακτέ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο τίμημα. Βοηθάει το βίο καθεστώς στο, στη βιότητά του και δεν αποτελεί μεγάλη πολιτική χειρονομία. Εγώ είμαι υπέρ αναβολής της ψηφοφορίας, αλλά ας ακούσουμε αυτά που μας είπε ο κύριος Γκάλερ. Ας δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες και ποιες θα ήταν οι συνέπειες για τα λιευτικά αποθέματα αν οι λιευτικοί πόροι πολιθούν σε χώρες που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη συντήρηση των ελευτικών πόρων και στις δικές ελευτικές συμφωνίες δεν εντάσσουν ρήτρε που βάζουμε στις δικές μας. Θα κλείσω το συζήτηση με τη δική μου παρέμβαση. Όλους σας άκουσα. Θα πρέπει να γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελευθερική Συμφωνία. Αύριο ή τέλο πάντων όποτε να είναι ανάλογα με το τι θα προτείνετε, να ληφθεί μία απόφαση. Να γίνει η ψήφιση και η ψηφοφορία, διότι έχουμε δεσμευτεί, πρόκειται για μία μακρά διαδικασία. Δεν είναι χτεσινό αυτό το θέμα εδώ και πολλούς μήνες. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδρομή και υπάρχει αυτή η δέσμευση. Και επομένω, κατά συνέπεια, έχουμε την επόμενη φάση. Δηλαδή, θα δώσει το πράσινο φω στο Συμβούλιο για την Ελευθερική Συμφωνία. Όμω, ήδη είναι δεδομένες κάποιες συμφωνίες, κάποιε υποσχέσει, Πάκτα σουν σερβάντα. Και στο τέλο Νοεμβρία, εάν δεν ε, κλειστεί αυτή η συμφωνία, τότε και εμεί θα έχουμε σπάσει την υπόσχεσή μα. Θα έχουμε δει την υπόσχεσή μα που την έχουμε δώσει. Και ο κλάδο θα έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Άρα, εάν ενεργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, πρόκειται να παραβλάψουμε τα συμφέροντα του κλάδου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή η ελληνική συμφωνία που είναι κάτι το οποίο ήδη εξηγήθηκε προβλέπει κάποιες ρήτρε και στο σώμα της συμφωνία και στο πρωτόκολλο. Οπότε σε περίπτωση που επιβάλλει κάποιες κυρώσει η Ένωση το Νοέμβριο ή και παραπέρα παραπέρα άπαξ και το Συμβουλίο εγκρίνει τη συμφωνία συντρέχουν λοιπόν στο 6 και στο 7 στις αυτές τις σχετικές ε, διατάξεις του πρωτοκόλλου ή του συμφωνίου προβλέπονται από λοιπόν αυτές οι ρήτρες που λένε ότι εάν πέσουν αυτές οι ρήτρες έχουμε αναστολή ισχύω της συμφωνίας. Άρα να πώς μπορεί να πληθούν κάποιες κυρώσεις τυχούνια η όσα έγιναν ή όσα μπορεί να πως μπορει να πληθουν καποιες κυρωσεις στιγμή οι μέχρι τις εκλογές. Προβλέπετε μας κάποια διαδικασία ούτω ώστε να γίνει αναστολή των πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σας λέω. Τώρα, μια που και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε την επόμενη φάση, δηλαδή την έγκριση στην Ολομέλεια. Κοιτάξτε θα κάνετε για να αποφασίσουμε αύριο. Θα έχετε ενημερωθεί και μπορούμε να προχωρήσουμε προς την επιλογή της ψηφοφορίας. Εάν τον Νοέμβριο έχουμε εξελίξεις που συντρέχουν προς τούτο, θα πάμε σε αναστολή των πληρωμών. Δεν πρέπει η Κομισιόν και το Κοινοβουλίο εμάς να κατηγορήσουν ότι μόνο εμείς προκαλέσαμε την αθέτηση των υποσχέσεών μας. Και ότι έτσι δεν χρησιμοποίησαμε το πιο πρόσφορο μέσο για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα για τα δικά μα και των άλλων. Άρα, αναβολή μέχρι αύριο όσον αφορά την ψηφοφορία τη ε, συμφωνία και εάν αύριο προκύψει κάτι άλλο, είδομε. Σα επαναλαμβάνω, υπάρχουν λύσει που μπορεί να, να, να χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Άρα, παρακαλώ και σας ζητώ να το αφήσουμε για αύριο το θέμα. Πάμε παρακάτω στο μέρος για που είναι το σημείο υπαριθμών 5. Αφορά την παρουσίαση τη γραμματέία του κυρίου Ολιβάρε, δηλαδή, που είναι ο διευθυντή της ΥΠΟΛ Β σχετικά με τι Υπηρεσίε θεματικού τμήματο. κάτι που γιατί τι προάλλε το είχαμε ξανασυζητήσει. Οπότε, και συζητήθηκε τι προάλλε, μια που οι περισσότεροι εδώ πέρα είναι καινούργοι θα το βρουν ενδιαφέρον να τα ξαναπούμε και γι' αυτό το βάλουμε στην αίσθηση και άρα ο κ. Ολιβάρες να σας εξηγήσει τι δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά το θεματικό αυτό τμήμα. Κύριε Ολιβάρες, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τι καλά που έχουμε αυτή την ευκαιρία να μπορέσω να σας παρουσιάσω τις, θεματικέ υπηρεσίε αυτέ υπηρεσίες αυτές όσον αφορά την αρρωγή προς τους κοινοβουλευτικούς για ε, αυτές τις υπηρεσίες, τις ερευνητικές γενικές γραμματείες του Κοινοβουλίου. Κάτι το οποίο προσφέρεται εις τα όργανα του Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Στα γαλλικά. Το 2004 αποφασίσαμε να διαρθρώσουμε τις υπηρεσίες της έρευνας, ούτως ώστε η έρευνα των ανεξαρτήτων γενικών διευθύνσεων τώρα να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας των βουλευτών, δηλαδή στις υπηρεσίες εσωτερικής ψηφίας πολιτικής. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε καλύτερη, μεγαλύτερη προσέγγιση και έτσι θα είχαμε τεχνική αρρωγή άμεση στους βουλευτές στα πλαίσια των συνήθων εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτή η υπηρεσία λέγεται θεματικό τμήμα. Η βασική μας αποστολή είναι να σας δίνουμε όποτε το ζητάτε, την εμπειρογνωμοσύνη μας, ούτως ώστε να επιτελείται το νομοθετικό σας έργο. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα να ποιε είναι οι τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά την νομοθετική δραστηριότητα, γιατί ο κόσμος μας είναι τόσο περίπλοκος βάζει οικονομικής, νομικής, τεχνολογικής, που εδώ και χρόνια δεν μπορέσουμε να αποφασίσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την νομοθεσία κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχει τέτοιου είδου βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη. Επίση, κάτι άλλο που αποφασίστηκε είναι να υπάρχει ένα ειδικό κονδύλιο στον προπολογισμό για την χρηματοδότηση των σχετικών μελετών γιατί έπρεπε να προσφύγουμε σε κάποιες ομάδες εμπειρογνωμόνων, σε κάποια ειδικά εξειδικευμένα ιδρύματα για να βοηθήσουν σε αυτές τις κοινωνικές δραστηριότητε. Οπότε και αυτές οι ερευνητικέ κινήσεις αφορούν πάλι αυτό το θεματικό τμήμα που λειτουργεί παράλληλα με την γραμματεία των Επιτροπών. Ο κύριος Φιλίπ Μουσκάρ είναι ο προστάμενος καθημερινά συνεργάζονται μαζί σας και επίσης έχουμε και τα θεματικά τμήματα από όπου προκύπτουν αυτά τα κείμενα εμπειρογνωμοσύνης για βοήθεια της κοινοβουλευτικής ε, εργασίας, για περιφερειακή πολιτική, για μεταφορές, για πολιτισμό, για, για αλία, δηλαδή οι βασικές ε, διαρθρωτικές πολιτικές που μας απασχολούν στο Κοινοβούλιο. Αυτές οι ερευνητικέ και διαχειριστικές ε, ενέργειες, ο τεχνοκρατικής, οικονομικής, που αφορούν εξωτερικές υπηρεσίες, πάλι πάγοντα το θεματικό τμήμα και εγώ ως διευθυντής έχω ως ε, καθήκον να προσέχω τόσο ώστε να υπάρχει στενή συνεργασία, άμεση στήριξη, κατόπιν φυσικά αίτηση των βουλευτών. Κάτι άλλο φαίνεται. Αυτό είναι το ότι δεν μιλάμε εδώ πέρα για κείμενα πολιτικά. Είναι τα κείμενά μας επιστημονική ανάλυση. Έχουμε και σύστημα ποιοτικού ελέγχου, ελέγχου της μεθοδολογίας της εργασίας μας, οπότε αυτό το πιθανό κάνουμε να στηρίξουμε τις κοινοβουλικές συζητήσεις. Και τελικά αποδεικνύεται το αν αξίζει η μελέτη μας από την ποιότητα της συζήτησης που ακολουθεί κατά τις κοινωνικές εργασίες κάποιες επιτροπές όπως η δική σας. Άρα σε εσά απόκειται να κανονίσετε το με τι θα ασχοληθεί η έρευνά μας. Τι μπορεί να σας βοηθήσει στις εργασίες σας. Εσείς δεν καθόσατε τα αντικείμενα. Και εσείς επίσης θα κανονίσετε πότε θα παρουσιάσουμε τις ε, μελέτες μας. Ε, ανάλογα με το αν υπάρχει Φερρυπίν ε, κάποια έκθεση, κάποια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Εμείς ως διοίκηση του Κοινοβουλίου θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, τεχνοκρατική, τεχνική αρτιότητα της δουλειάς σας. Να υπάρχει κάποιο ανεξαρτησία των όσων σας παρέχουμε σαν βοήθεια. Όσον αφορά την επιστημονική πτυχή των θεμάτων πρέπει να συζητήσετε και επίσης αναβάλουμε και την ε, ευθύνη όσον αφορά κάποιες συμβάσεις, κάποιες αναθέσεις εξωτερικούς συμβούλους. Επίσης έχω την αρμοδιότητα για την χρηματοδότηση των σχετικών μελετών. Και έχω την αρμοδιότητα της ε, προστασίας των οικονομικών συμφωνών του Κοινοβουλίου. Με δύο λόγια αυτά θα να σας πω. Αλλά τώρα τη σκητάλη θα πάρει ο συνεργάτης μου Χεσούς Ιμπόρα. Που ασχολείται πιο ειδικά με την ε, αλλή, οπότε θα σας πει ακριβώς ποιες είναι οι λεπτομέρειες του συστήματος. Και κατόπιν έχουμε τον κύριο Λιβέρα Γκόμες που είναι οι τμήματάρχες του θεματικού τμήματος. Και αυτή θα σας εξηγήσει πώς και τι να ζητάτε και ποια είναι τα πλαίσια μας, τα οικονομικά στο οποία κινούμαστε. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, δώστε το λόγο στον κύριο Μπόρ για να σας εξηγήσει. Έχετε το λόγο. Muchas gracias, Να σα πω τι λεπτομέρειε τη λειτουργία του, τμήματό μα. Το 2004 ξεκινήσαμε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να σα δώσουμε από τεχνοκρατική πλευρά και επιστημονική πλευρά βοήθεια κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει, σταμάτησε ο μιλητή. Fueron creados en 2004 para suministrar asesoramiento. Και έτσι παργίνεται η αξιολόγηση. Και έτσι έχουμε κάποια στοιχεία για να βοηθηθεί το κοινωνιστικό έργο. Και ακριβώ ε, μπλεκόμαστε στο έργο σα, ακριβώ όπω σα τα εξήγησε ο κύριο Ολιβάρη. Τα θεματικά αυτά τμήματα έχουν κάποιο είδου ε, ε, προπολογισμό. Και επίση πρέπει να προσέχουμε να προστατεύουμε τα συμφέροντα τη κοινότητα. να τηρούμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό και με αυτό ασχολούνται οι διευθυντές και οι γενικοί διευθυντές. Στις ιστορικές πολιτικές έχουμε τέσσερα θεματικά τμήματα. Το ένα είναι συνοχή, διορθωτικές πολιτικές, καλύπτει πέντε τομείς. Γεωργία, πολιτισμός, αλληλεία, περιφερειακή πολιτική και μεταφορές. εξωτερικέ εξωτερικές πολιτικές έχουμε μόνο ένα θεματικό τμήμα από την άλλη μεριά. Παρακολουθούμε από κοντά τις εργασίες τη Επιτροπής. Έχουμε στενή συνεργασία και γίνεται αξιολόγηση ανεξάρτητη. Τώρα η οργάνωση αυτών των θεματικών λιμάτων γίνεται ανάλογα με τι ανάγκε και το τι θα ζητήσουν οι επιτροπέ, όμω έχουμε το προσωπικό του Γενικού Γραμματέα, ε, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να ζητήσουν βοήθεια, όπω και οι διευθυντέ και οι γενικοί διευθυντέ. Το 2008 ε, είχαμε και αναθέσει προ εξωτερικού συμβούλου. Φτάσαμε στα έξοδα των 8 εκατομμυρίων ευρώ σαν, σαν πρικοδότηση και τελικά ξοδέψαμε τα 7. Το 2009 είπαμε ότι η δραστηριότητα ε, θα είναι διαφορετική λόγω των εκλογών. Αυτά που ισχύουν και για την εξέλιξη του τομέα της Ελίας, γιατί υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με την αύξηση της ζήτησης ανθρώπινου πόρου σε σχέση με την πρικοδότηση που είχαμε. Το 2009 επομένω είναι μια ειδική, ξεχωριστή χρονιά, γιατί μέχρι το τέλος του 2009 δυστυχώς στις διαφάνειες δεν μπορεί να δείτε αυτά τα στοιχεία. μέχρι το τέλος του 2009 θα έχουμε περί τα 44.000 ευρώ και λόγω των διαδικασιών που προβλέπονται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε αυτά είναι το να έχουμε ε, κάποια ενημερωτικά εσωτερικά σημειώματα. Η αξιολόγηση του θεματικού τμήματος γίνεται εσωτερικά από τους, το προσωπικό του κοινοβουλίου και ε, αν χρειαστεί μπορεί να προσφύγουμε και σε εξωτερική αξιολόγηση. Αυτό γίνεται με διαδικασίες διαγωνισμών και ανάθεση. Ξεκινά αυτή η διαδικασία αιτήση της Επιτροπής Αλίας μέσω του συντονιστή και έτσι έχουμε απόφαση των συντονιστών, την εγκρίνουν η Επιτροπή και κατεβαίνει σαν αίτημα όλης της Επιτροπής έχουμε ως προϊόντα στα θεματικά τμήματα διάφορα θέματα. Έχουμε κάποια εργαστήρια, τα λέμε, workshop. Έχουμε τις εσωτερικά σημειώματα και έτσι μπορούμε να συμπληρώσουμε τη δική σας δουλειά ή ακόμα και να αντιτάξουμε κάτι σε αυτό το οποίο λέτε. Να σας διορθώσουμε δηλαδή. Βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια τι γίνεται με τα υπόλοιπα προϊόντα του συνόλου των θεματικών τμήματων. Είναι λίγο διαφορετικά όμω τα πράγματα στην Ελία. Βλέπετε ότι χρειάζονται περισσότερα ιστορικά σημεία και ιστορικέ μελέτε. Εδώ βλέπετε τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, περισσότερες μελέτες εις βάθος για τις διάφορες νομοθετικές διαδικασίες. πρόθεσμα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις νέες ανάγκες της Επιτροπής Αιλίας στα πλαίσια της συναπόφασης. Άπαξ βέβαια και εγκριθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο στόχος του θεματικού τμήματος είναι το να έχουμε ξεκάθαρα αξιόπιστα έγγραφα που να βοηθάνε τις εργασίες σας. Είναι μέσα αποτελεσματική αλλά και Γρήγορη, θα πρέπει το αντικείμενο του αιτήματο αλλά και το περιεχόμενο να μα το ξεκαθαρίζεται όσο γίνεται με πιο μεγάλη ακρίβεια. Εξωτερική ανάθεση γίνεται συνήθω το τέταρτο τρίμηνο. Σε συνέχεια μελετών τη προηγούμενη χρονιά. Οπότε και εκεί πέρα, όσο καλύτερα προετοιμαστεί κανεί, είναι πιο, πιο ποιητικό το προϊόν. Δύο πάρα πολύ βασικά ζητήματα αυτής της ε, θητείας είναι η μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ και η μεταρρύθμιση στις κοινέ οργανώσεις αγοράς. Βλέπετε εδώ και άλλες μελέτες που έχουν γίνει, που γίνονται και αφορούν αυτές τις, αυτά τα θέματα. Μεγάλη είναι η ζήτηση επομένως για αυτές τις μελέτες. Επίσης, θα γίνουν και άλλες τρεις μελέτες όσον αφορά την ε, στρατηγική για την βιώσιμη ηχθειοκαλλιέργεια. Και αυτές θα αφορούν βέβαια τη δουλειά της Επιτροπής Ελίας. Θα μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη ή σε κάποιες ε, προθήκες του τρίτου, του τρίτου και στο website της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών ή γενικότερα στο website του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί που λέει activities παρακάτω πάει ε, επιτροπές και παρακάτω μελέτες. Έχουμε αυτό το newsletter και μπορείτε να δείτε ε, πότε προκύπτουν κάποια καινούργια προϊόντα. Για ό,τι θέλετε, στείλτε μας ένα email. Eh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ολιβέρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Για να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση που υπήρξε λεπτομερέστατη, θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω κάποια θέματα. Λοιπόν, έχουμε μονάδες έρευνας και αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία όσον αφορά τι δημοσιονομικέ δραστηριότητε. Συγγνώμη, νομοθετικέ δραστηριότητε των κοινοβουλευτικών επιτροπών, διορθώνει η ομιλήτρια. Κάναμε πάρα πολλέ έρευνε, εκατοντάδε έρευνε ε, κατόπιν αιτήματο ε, των διαφόρων ε, βουλευτικών επιτροπών των αρμοδίων. 123 μελέτες ετοιμάσαμε, 161 εσωτερικά σημειώματα, 52 briefing papers, ε, με εργαστήρια για την Επιτροπή Αλλιές 19 μελέτες, 34 εσωτερικά σημειώματα, 19 briefing papers, 4 εργαστήρια. Χωρίς να μιλήσουμε για τα διάφορα τεχνικά δελτία που ετοιμάζουμε συχνά. το, τμήμα στο θεματικό συνεργάζεται στενά με την γραμματεία της Επιτροπής Αλλιές και όπως αναφέρθηκε υπογραμμίζω ότι μέχρι τώρα μόνο ένας υπάλληλο την υπεύθυνο για την αλία στο θεματικό τμήμα. Ευτυχώς, μια νέα συνάδελφο, η κυρία Μπομπέσκο, που κάθεται εκεί πίσω, ήρθε να μας ενισχύσει. Προσέξτε και το θέμα του προπολογισμού που στη διάθεσή μέχρι το τέλο του 2009, περίπου 44.000 ευρώ. Όσον αφορά τον προπολογισμό η τεχνογνωσία 2010, πιθανότατα θα είναι τη ίδια τάξη μεγέθους όπω αυτός που είχα τη διάθεσή σας το 2008, 360.000 ευρώ περίπου. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό να υποβάλλετε αιτήματά σας για τεχνογνωσία για τις εκθέσεις που προβλέπετε το ταχύτερο δυνατόν. Κανονίστε τον συντονιστέ σας. Ή καλύτερα, όσο πιο νωρίς λάβουμε τα αιτήματά σας στο θεματικό τμήμα, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν τα δέοντα. άρα και θα είναι καλύτερη τελική ποιότητα των μελετών. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν ερώτημα που θα επιθυμούσατε να μου θέσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει ερώτηση. Έχετε ερώτηση για κάποιους από αυτούς που παρενέβησαν. Όχι. Ε. Por su claridad en sus exposiciones, dado que no han suscitado. Ah, sí, perdón, el señor Gallagher quiere hacer una pregunta. Just a quick question. We got a lot of Ένα γρήγορο ερώτημα. Έχουμε πολύτιμε πληροφορίες, αλλά θα είναι πολύτιμε αν έχουμε ένα αντίγραφο. Να έχουμε τις λεπτομέρειες με ονόματα, επαφές. Οι πληροφορίες ε, έφυγαν γρήγορα από την οθόνη. Πάμε στο στενά χαρτί, να μα στείλετε με διευθύνσει, ονόματα, εκείνου που μπορούμε να τους σε επαφή κλπ. Όσον αφορά τι παρουσιάσει, τυπώθηκαν και έπρεπε να διανεμηθούν και θα τα λάβετε. Pues eh, se repartirán eh, a lo largo de la, de la reunión. Cuando estén en... Sí, ya, ya se han repartido, están aquí. Sí, la tienen ustedes en sus... Δεν ξέρω όχι αν έχετε λάβει αυτό το έγγραφο, αν υπάρχει στους φακέλους σας. Σας ευχαριστώ για το όσο είπατε. Πάμε στο πολύ μας δίδεξη. Πρώτα απ' όλα δούμε το 6, γιατί ε, θα τα πούν οι συντονιστέ και θα μα ε, ενημερώσουν. Για μην υπάρχει όμω αύριο πρόβλημα. Στι 9 θα έρθει ο διευθυντή αρμόδιο για τι ελληνικέ συμφωνίε. οπότε μπορείτε να του θέσετε όλα τα θέματα. Οπότε να αναβάλουμε την ψήφιση και θα το δούμε στις 10 η ώρα ούτως ώστε όλοι οι βουλευτές και να το πείτε ξέρω τον εδώ ότι στις 10 ακριβώς θα αρχίσει η ψήφιση. Στις 10, στις 10 επομένως θα ψηφίσουμε σε σχέση με την Ελευθερική Συμφωνία. Πάμε τώρα στο έκτο σημείο της Μέσης Διατάξεως. Υπόγλωσσος στο πλαίσιο της οργάνωσης αλλήλειας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, ΝΑΦΟ. Τις προάλλες το συζητήσαμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα θα πρέπει να μεταφέρουν στο κοινωτικό δίκαιο αυτά τα οποία αποφασίστηκαν από τον ΝΑΦΟ το 2007. προσωρινά εφαρμόστηκαν με τους κανονισμούς που αφορούν τις ποσοστώσεις, τα ΤΑΚ, για το μέγιστο επιτρεπόμενο αλλήλεγμα. Και θα πρέπει με την νομοθετική διαδικασία να γίνει μεταφορά λοιπόν των διατάξεων όπως πρέπει στο κοινοτικό δίκαιο. Επαφές έγιναν με τον κλάδο και τελικά είναι σύντονη κάθε απόφαση, κάθε πρόταση της Κομισιόν με τις αποφάσεις αυτές. Οπότε πρέπει να εγκρίνουμε αυτό το, αυτή την πρόταση της Κομισιόν Και όπως έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να δούμε από ε, τον ΝΑΦΟ ή από τι άλλε περιφερειακέ οργανώσει, ό,τι απόφαση λαμβάνεται θα πρέπει να μεταφέρει στο για όσο γίνει πιο γρήγορα και με τι πιο σωστέ και δόκιμε διαδικασίε. Γιατί τελευταία, ε, λόγω ελλείψη ανθρωπίνων πόρων, έγινε η μεταφορά με άλλους τρόπους, με κανονισμούς τάξη και ποσοστώσεων. Αυτό ήθελα να σας πω. Τώρα έχουμε τον κύριο Νίλσεν. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να πει όσα άκουσε. Ε, πρώτα έχει το λόγο ο κύριο Νίλσεν και κατόπιν οι βουλευτές. Η κυρία Νίλσεν. Α, συγχωρήστε με. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι συνηθισμένη στο λάθος αυτό με το επίθετό μου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα προς το παρόν. Έριξα μια ματιά βέβαια στην έκθεση του εισηγητού. Ευχαριστούμε πολύ για τις διαδικασίες που έχει κινήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημειώνουμε και τα σχόλια που έγιναν σε ό,τι αφορά την άμεση μεταφορά στις, ε, των συστάσεων που γίνονται για τα ΝΑΦΟΣ. Ευχαριστώ. Nada que eh, anuncio que el plazo de presentación de Η προθεσμία της τροπολογίας είναι η 7η δεκάτου το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε 3 Νοεμβρίου στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, 7 δεκάτου για τις τροπολογίες το μεσημέρι. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Οπότε έτσι τελειώνουμε και με το σημείο 6 της μέση διάταξης. Και πάμε στο 7. Η συζήτηση που αφορά την πράσινη βίβλο για τη μεταρρύθμιση τη κοινή ελευθερική πολιτική. Κυρία Πατράου, είστε η συγγήτρια και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ την πρόεδρο, την κυρία Φράγκα, γιατί από την αρχή προωθούσε αυτή την πολυπόθητη μεταρρύθμιση του τομέα της αλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να συγχαρώ μάλλον την Επιτροπή, γιατί πραγματικά είναι πολύ σωστή χρονική στιγμή που υποβάλλεται αυτή η πράσινη βίβλος, ειδικά στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης που περνούμε. Γιατί δημιουργεί ακόμα ένα πρόβλημα για τον πρωτογενή τομέα. Ε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και τα μέλη και τους συντονιστές φυσικά. Τους ε, κοινωνικού εταίρου, όσου συνεργάστηκαν. Πραγματικά είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η σύμπνοια για την ε, βελτίωση του τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε κάποιες οδηγίες για την ε, μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική. Το δεύτερο μισό της ε, δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 είδαμε πραγματικά μία μείωση στους θαλασσίους πόρους και αυτό είχε ε, σημαντικές οικονομικές ε, επιπτώσεις. Μέχρι τότε η θάλασσα ήταν ε, μια πηγή αλληλείας χωρίς τέρμα. Η απώλεια όμως διαφόρων ειδών από τις παράκτιες περιοχές, από τις παράκτιες περιοχές μέχρι και την ανοιχτή θάλασσα, δεν οφείλεται σε νέες τεχνολογίες ή σε παρεμβατική ε, αλία. Απλώς ε, όλοι ε, οδηγούνται σε τέτοιες πρακτικές και όλο και περισσότεροι ανέφεραν παράπονα και προβλήματα λόγω ακριβώς αυτής της υπεραλίευσης. Το περιβάλλον επιβαρύνθηκε, Έγινε συγκέντρωση των αληφτικών προσπαθειών σε συγκεκριμένες περιοχές, ε, κλιματικές αλλαγές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πραγματικά αποτέλεσαν ε, παράγοντες ζωτικής σημασίας που πίεσαν ακόμη περισσότερο ε, και αύξησαν την μείωση των αληφτικών πόρων. Κάποια είδη που είχαν αρκετά σημαντικό πληθυσμό τώρα άρχισαν να εξαφανίζονται. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα ο τομέας της αλίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν μερικώς ή με τομεακή προσέγγιση. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη οριζόντια προσέγγιση, έτσι ώστε να δράσουμε προς όλα τα μέτωπα. Οι διασυνδέσεις που υπάρχουν είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να εκτιμηθούν αναλόγως. Όταν συζητούμε την ε, πράσινη βίβλο για τη θαλάσσια πολιτική, μπορούμε να εμπλέξουμε και εκεί την ε, αληφτική πολιτική. Δεν μπορούμε να έχουμε κατακριματισμένη προσέγγιση. Πρέπει να συνδυάσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να τα θέσουμε σε ένα γενικό πλαίσιο, να βρούμε ποια είναι η, ποια είναι η αιτία του προβλήματος και να βρούμε ε, αποτελεσματικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε όντως να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στον τομέα της αλληλείας, έτσι ώστε να έρθουμε και να υποβάλουμε ένα παράδειγμα το οποίο θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ειδών, την έλλειψη αλληλευτικών αποθεμάτων, την ε, επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφείς ορισμούς, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, εφόσον θέλουμε όντως να βοηθήσουμε τις ελευτικέ δραστηριότητες. Βρισκόμαστε βέβαια και εν το μέσο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που και αυτή επιβαρύνει την κατάσταση όχι μόνο στην λειτουργία και στην ανάπτυξη της αλληλείας ως ε, δραστηριότητας αλλά επιβαρύνεται η κατάσταση γιατί δεν υπάρχουν άλλες επιλογές για τους αλληλείς. Δεν μπορούν να βγάλουν το ψωμί τους διαφορετικά τα τάκ οι ποσοστώσεις δεν θα βοηθήσουν ε, στην αύξηση της παραγωγής ή δεν θα τους δώσουν τα περισσότερα έσοδα από την αύξηση της παραγωγής. Επίσης υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται και στην, ε, στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης ε, επιβαρύνεται ο τομέας της αλληλείας, τα αποθέματα, η θερμοκρασία αυξάνεται, η η όξυνση των θαλασσών, όλα αυτά είναι τομείς που επηρεάζουν πραγματικά το, ε, τις θάλασσες και όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει να αντιμετωπιστούν η ε, διακύμανση των τιμών του πετρελαίου επίσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που με τον τρόπο τους συμβάλλουν και έτσι είναι δύσκολο για όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό να έχουν ένα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Οι τιμές επίσης ε, είναι πολύ χαμηλές για τους αλληλείς, οι τιμές των ε, αλλιευμάτων. Μπορεί να ε, τους επιβληθούν κυρώσεις για παραβάσεις. Μερικές φορές δεν υπάρχουν όμως και αρκετά αλλιεύματα για να ψαρέψουν. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος στόλος ευρωπαϊκός και υπάρχουν και δυσκολίες στην παροχή αλλιευμάτων προς την ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, η υδατοκαλλιέργεια ε, αυξάνεται. Ε, πώς λοιπόν μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ε, τα σχέδια που υιοθετούμε κυρίως είναι βραχυπρόθεσμο όχι μακροπρόθεσμο Πώς λοιπόν μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα για τον αληφτικό τομέα. Πρέπει να τα ορίσουμε όλα αυτά σαφώς, έτσι ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν, τι αποφάσεις πρέπει να λάβουν, πού θα βρούμε τα λεφτά πώς μπορούμε να ε, επενδύσουμε στους, σε σωστές δραστηριότητες και όχι σε δραστηριότητες που τελικά δεν ε, μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα. Επίσης, έλλειψη εμπλοκής, συμμετοχής των ε, φορέων που εμπλέκονται στην όλη δραστηριότητα της αλληλείας. Και σε αυτό είχαμε πρόβλημα. Πολύ συχνά δεν ε, βασιζόμαστε, δεν χρησιμοποιούμε τη γνώση που έχουν οι ίδιοι αλληλείς για την περιοχή στην οποία αλλιεύουν. Την πρακτική γνώση πολλές φορές θα ήθελαν οι ίδιοι οι αλληλείς να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους ε, περιφέρεια για τη δική τους περιοχή αλίευσης. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, γιατί δεν τους λαμβάνουμε υπόψη, γιατί δεν δημιουργούμε ώστε να μειωθεί επίσης η έλλειψη συμμόρφωσης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μια γενική ε, δραστηριότητα, μια γενική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε τα βασικά προβλήματα. Ε, εγώ αυτά ε, θεωρώ στα πιο σημαντικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν γενικές αρχές για να δομήσουμε σωστά τον τρόπο με τον οποίο θα επέμβουμε στον τομέα της αλίας. Πρέπει, όπως είπα, να, να προστατεύσουμε, να διατηρήσουμε τα αποθέματα ε, τα αλλιευτικά. Να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο εισοδημάτων ε, για τους αλληλείς, έτσι ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια, να διατηρήσουμε την ε, αλληλεία. Ας χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλληλείας ως ε, απόφθεγμα όλων αυτών των προσπαθειών. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον πληθυσμό των ε, ειδών τα αποθέματα με βιώσιμο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν οι αλληλείς να συνεχίσουν τις δραστηριότητε τους. Αυτές νομίζω είναι οι βασικές προτεραιότητες, οι βασικοί στόχοι της αλληλευτικής πολιτικής. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Μιλούμε για την εναρμόνιση ε, των, ε, όλων των εμπλεκομένων φορέων και των συμφερόντων τους. Πρέπει να εκπονήσουμε να δημιουργήσουμε έτσι μια νοοτροπία ε, σύμφωνα με την οποία οι κανόνες τηρούνται. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανάληψη ευθύνης που έχει επίσης να κάνει με την εφαρμογή των μέτρων στα κρατη Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε με ευελιξία. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς αυτό. Επίσης, η διαχείριση της ε, αλίας, πολύ σημαντικό για τους ε, υπουργούς, γιατί αυτή είναι που θα πάρουν βέβαια την τελική απόφαση. Η διαχείριση όμως της ε, αλλήλία θα πρέπει να έχει μια πιο έντονη πτυχή ε, περιφερειακή. Πρέπει να ενισχύσουμε τις, ε, τα συμβούλια, τα περιφερειακά ή τις συνελεύσεις τις περιφερειακές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμβολή από τους επιτόπου ανθρώπους. Επίσης να τους εμπλέξουμε περισσότερο, να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, όχι απλώ να τους λέμε τι να κάνουν, έτσι ώστε το σύστημα διαχείρισης να βασίζεται σε αυτό που ξέρουν οι άνθρωποι εκεί, όχι απλώ να τους λέμε τακτή και να είμαστε πιο ε, ευέλικτοι και λιγότερο γραφειοκρατικοί και να είμαστε πιο κοντά στου ίδιου του αλληλεί. Άλλη μια πρωτοβουλία που επίση θεωρώ ότι είναι ε, σημαντική και για την οποία επίση εξευρέθη συνένεση ήταν η οριζόντια φύση των δραστηριοτήτων μας. Προσπαθούμε όντω να ανθίσει οικονομικά ο τομέας μέσω χρηστής διαχείρισης των πόρων. Προσπαθούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη βιώσιμη απόδοση του τομέα. Και κάτι άλλο επί του οποίου μάλλον θα συμφωνήσουμε είναι ότι ο τομέας της αλληλείας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Επίσης θεωρώ ότι συμφωνούμε επί των αρχών που διέπουν τον τομέα αυτό και πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν καμιά φορά αμφιλεγόμενα και επί των οποίων κάποιοι συμφωνούν και κάποιοι όχι. Σε αυτό το τομέα λοιπόν ε, υπάρχουν κάποιοι μανατομίες που όντω μπορεί να είναι αμφιλεγόμενοι και να δημιουργήσουν προβλήματα. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητοι. τι μπορούμε να κάνουμε για, τις, για τη δυνατότητα ελίευσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ποια μέτρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να αναλάβει ο τομέας την ευθύνη που του αναλογεί. Όταν δείτε την πολιτική, μιλούμε για μια διαχείριση που βασίζεται σε αποτελέσματα. Οι δημόσιες αρχές θέτουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί ο κλάδος. Βέβαια, εντάξει, δίνεται και ένα περιθώριο λιγμών, οπότε τα περισσότερα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι ε, τομείς που πρέπει να συζητηθούν και ένας από αυτούς είναι η εγγύηση της παράκτειας αλληλείας η εξασφάλιση της ε, παράκτης Αυτό θα πρέπει ίσως να το δούμε με λίγο πιο διαφορετικό τρόπο στα πλαίσια της ΚΑΠ, γιατί μιλούμε και για μέτρα για βιο, τους βιομηχανικούς στόλους. Οπότε αυτό πρέπει να το δούμε επί τη βάση της οικονομικής αποδοτικότητας. Όταν μιλούμε πάλι για μικρού επίπεδου ε, αλία, για αλία δηλαδή μικρών κοινοτήτων, ίσως εκεί πρέπει να δούμε περισσότερο την κοινωνική πτυχή των πραγμάτων. Άλλο ένα τομέα που πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα είναι η ενσωμάτωση της ΚΑΠ σε ένα πιο ευρύ ε, πλαίσιο θαλασσιών πολιτικών. Εδώ πρέπει να πούμε πως η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να εγγυάται μία προσέγγιση προς το θαλάσσιο περιβάλλον που θα βασίζεται στα οικοσυστήματα. Υπάρχει και η σχετική ε, οδηγία πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη την πτυχή του περιβάλλοντος όταν μιλούμε για τέτοιες καταστάσεις. Ένταξη λοιπόν της ΚΑΠ στην πολιτική, στη θαλάσσια πολιτική. Για να γίνει αυτό πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε τη γενίκευση των προβλημάτων σε ό,τι αφορά τον τομέα της αλίας και πώς επίσης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Και αυτό είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή πολιτική της θάλασσας η ΚΑΠ στο μέλλον θα πρέπει να ενταχθεί στις, σε αυτές τις ε, πολιτικές και ειδικά στη θαλάσσια πολιτική. Επίσης, πρέπει να δοθεί η απαραίτητη σημασία στην, ε, στην με συγκεκριμένη στρατηγική, καλύτερη και ε, πιο αποτελεσματική ε, χρήση των ε, διαδικασιών, ε, ταχείες διαδικασίες, έτσι ώστε να καταλήγουμε σε αποτελέσματα πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά μεμονωμένα σημεία τα οποία πρέπει να δούμε. Δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω, γιατί ούτως ή άλλως είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε, αλλά θα ήθελα απλώς να πω, αν δείτε τις διατάξεις της πράσινης βίβλου και το χρονοδιάγραμμα, 30 Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου λέει θα γίνει πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα δηλαδή. Μετά 3-4 Νοέμβρη δεύτερη συζήτηση. Ίσως θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε και κάποιους ε, για να συζητήσουμε μαζί τους. Θα, ε, επίσης μετά θα λάβουμε την ε, έκθεση της Κομισιόν και αρχές Δεκεμβρίου Πρώτη ακρόαση 27-28 στην Επιτροπή μας α, ε, ψηφοφορία ε, το Γενάρη και 24 Φλεβάρι στην ε, Ολομέλεια. Αυτό το χρονοδιάγραμμα όμως μπορεί να αλλάξει και κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει. Ειδικά όταν ε, γίνει και η ακρόαση Οπότε θα ήθελα να μου επιβεβαιώσει αυτό το χρονοδιάγραμμα η, γραμματεία. Γιατί αν δεν μπορεί να τηρηθεί, ίσως να πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Βάζοντας ήδη ε, στο πρόγραμμα και τις διάφορες ακροάσεις στην, ε, στις επιτροπές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να, να εντάξουμε και την ε, διαδικασία που αφορά την πράσινη βίβλο όλη αυτή τη διαδικασία μελέτης της ε, ΚΑΠ. Επίσης ζητώ από τους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν να μην προχωρήσουν χωρίς τη δική μας γνώμη. Φαντάζομαι ότι και η δική μας άποψη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Πράσινης Βίβλου. Ευχαριστώ. Eh, Πρώτα να δώσω λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν στους βουλευτές. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Χαίρομαι που η κυρία Νέβες, η συγκήτριά σας, συμμερίζεται την ανάλυση μας και θεωρεί σκόπιμη τη μεταρρύθμιση. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν το συμμερίζονται όλοι σήμερα. Είναι ένα πρώτο σημείο που με ικανοποιεί. Ξέρω ότι οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βασίζονται σε κοινή αντίληψη περισκοπιμότητας της προσπάθειας. Θα ήθελα να πω μετά ότι στα εντοπιστέντα προβλήματα, αυτά που ανέφερε η κυρία αναγνωρίζουμε και τις παρατηρήσεις και τις Κομισιόν που έγιναν στην Πράσινη Βίβλο και τα ερωτήματα που ετέθησαν για τις λύσεις ε, αναφέρονται εκτενώς στην Πράσινη Βίβλο. Έχουμε μια απαρχή κοινή αναλύσεως, η οποία θα πρέπει να μας οδηγήσει η ανάλυση σε αυτή προς κοινή προσπάθεια. Και προτείνουμε στην κυρία Νέβες να εργαστούμε αν το θέλει και αν θέλει και άλλες πληροφορίες να της δώσουμε πληροφορίες. Για το χρονοδιάγραμμα υπάρχει κάτι σημαντικό που έθεσε η κυρία Νέβες. Οι εργασίες της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να ολοκληρωθούν πριν η Ολομέλη του Κοινοβουλίου ή η Επιτροπή προβούν σε ανάλυση της ε, ανακοινώσεως. Αυτό το σημειώνω. Eh, eh, eh, Ευχαριστώ. Ρομέβα. Ο κύριος Ρομέβα. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Για να δούμε επομένω. Υπάρχουν κάποια σημεία που ενδεχομένω είναι για το μέλλον σημαντικά. Τέσσερα. Εγώ έχω επισημάνει. Είμαι εισηγητής όσον αφορά τον ελεγκτικό κανονισμό και μπόρεσα να επισημάνω ποια είναι τα θέματα των ελεγκτικών μηχανισμών. Να έχουμε επικάλυψη, να έχουμε συντονισμό μεταξύ των δύο διαδικασιών. Συντονισμός όμως και όχι επικάλυψη. Και ένα από τα βασικά προβλήματα του ελέγχου είναι το ποιε είναι ακριβώ οι αρμοδιότητε τη ε, Κομισιόν. Έχει αρμοδιότητα να ασκεί το σχετικό έλεγχο η Κομισιόν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ό,τι κάποια να έχουμε θα πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς δυνατότητα εφαρμογής των ελεγχτικών κανονισμών τότε οι νόμοι μένουν νεκρό γράμμα. Αυτό πρώτο στοιχείο. Δεύτερο, να έχουμε κάποια συνέπεια. Κάτι το οποίο απασχολεί και και τον κόσμο σήμερα, δηλαδή το πώ χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι πόροι. Είναι ταυτόχρονα και παράδοξο. Είναι ταυτόχρονα και αιτία μεταρρύθμιση του ότι πολλέ φορές έχουμε την υπεραλίευση που χρηματοδοτήθηκε από τον δημόσιο κοργανό. και επίσης δύσκολα να εξηγήσει κανείς στον φορολογούμενο ή στον ψηφοφόρο ότι τώρα θα πρέπει να βάλουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη ούτως ώστε να περικόψουμε τους αλληλευτικούς στόλους εκείνους που προηγουμένως τους στηρίζαμε. Άρα, αυτά είναι πολύ σημαντικά από πλευρά πολιτική για αυτή τη μεταρρύθμιση και να κάτσουμε να βρούμε ποιος φταίει για τα προβλήματα αυτά. Επομένως, να μην πληρώνει την ύφη το λάθος πρόσωπο, να δούμε ποιος θα ωφεληθεί από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Να δούμε τι θα γίνει με την παραδοσιακή αλία. Εκεί έχουμε τρόπο αύξηση της απασχόλησης αλλά να κάτσουμε και να νομοθετήσουμε λαμβάνοντας υπόψη και το περιβάλλον και τις κοινωνικέ συνθήκες και τις συγκεκριμένες συνθήκες του τόπου όπου ασκείται η κάθε τέτοια δραστηριότητα. Και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Ε, και επίσης εδώ πέρα υπάρχουν δυνατότητε, πάρα πολύ σημαντικέ να αναπτυχθούν επίσης κάτι άλλο σχετικά με την ηχθειοκαλλιέργεια. δεν είμαστε και τόσο φανατικοί οπαδοί, αλλά το σημαντικό είναι να μην ξεχνούμε ποια είναι τα όρια. Περιορισμοί που πρέπει να έχει με τέτοια δραστηριότητα. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει έλεγχος του μέχρι πού μπορεί να φτάσει η επέκταση της δραστηριότητας. Θα πρέπει να ξέρουμε επίσης πού θα πρέπει να έχουμε ηχθειοκαλλιέργειες και πού όχι. Έχουμε κάποιες περιοχές, της Νατούρα, Natura, άλλες προστατευόμενες. Προσοχή, γιατί αν δεν το φροντίσουμε αυτό θα στείλουμε πολύ λάθος σήμα. Και στη Γαλλική υπάρχει πρόβλημα. Άρα αυτό θα πρέπει να το πούμε να διαπνέει κάθε πολιτική βοήθεια προς την ε, ηχθειοκαλλιέργεια. Yo de todas pediría que los temas de acuicultura se van a tratar a continuación. Πρόεδρος. Μετά θα τα πούμε τα συγκεκριμένα. με άλλη έκθεση. Για να ε, συγκεντρωθούμε τώρα στα δύο θέματα των εισηγητών που τώρα μας αποσχολούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για πολύ καλή αρχική παρουσίαση. Όσον αφορά τη συζήτηση που προηγήθηκε με τον κύριο Λιβάρας, μήπως χρειαζόμαστε πολλές λεπτομέρειες, λεπτομερή εξέταση, κυρίως των νομικών συνεπειών που συνεπάγονται, που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση της αληθικής πολιτικής. Μιλάμε για αλλαγή του φόρου, του συστήματος ποσοστώσεων. Πάμε σε ένα σύστημα η ITQ ή προσπάθεια που θα βασίζεται, η προσέγγιση βασίζεται μόνο στην προσπάθεια ή μείγμα ποσοστώσεων, προσπάθειας όπως την πελαγική ε, αλία, πελαγική αλία μπορούμε να κρατήσουμε το σκουβό, να κρατήσουμε τα ITQ. Μπορεί να βασίζεται το σύστημα στην προσπάθεια, στην ρευτική προσπάθεια, που είναι καλύτερο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε νέες προσεγγίσεις. Επίτροπος αναφέρθηκε στο πώς μπορούμε να μεταφέρουμε την αξία, την ποσόστοση που έχουν ήδη οι στην αξία των ημερών στη θάλασσα Υπάρχουν νομικές επιπλοκές προς εξέταση. Και πώς μπορούμε να παγιώσουμε σχετική σταθερότητα σε ένα ενδεχόμενο σύστημα, αν αλλάξουμε από φόρους και ποσοστώσεις, σε ένα σύστημα που μετράμε τις μέρες στη θάλασσα. Μπορούμε να προστατεύσουμε τους αλληλείς με παραδοσιακά δικαιώματα αλληλεία σε συγκεκριμένη ζώνη. Πώς Μήπως πρέπει να ζητήσουμε νομική συμβουλή να εξεταστούν τα ITQs οι μέρες στη θάλασσα και να δούμε πώς θα μεταφερθούν διάφορα δικαιώματα από το ένα σύστημα στο άλλο και πώς μπορεί να επιληθεί σχετική σταθερότηση. Και μήπως η τρία έχει ετοιμάσει κάτι που είναι ειδική για το θέμα, έχει κάτι να προτείνει. Ποιε είναι οι απόψει. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Άντοτς. Τρία Τον Απρίλιο, όταν ξεκίνησε η Πράσινη Βίβλος, εκδόθηκε η Πράσινη Βίβλος, πολλοί ψαλάδες από την περιοχή μου, από την ε, Βόρεια Ιρλανδία, έβγαλαν στεναγμό ανακούφισης. Είπαν επιτέλους, βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Από μπορεί να γλιτώσουμε τους γραφειοκοτικούς ελέγχους. Η κοινή ελευτική πολιτική έχει αποδεκατήσει τον ελευτικό τομέα στη Βόρεια Ιρλανδία. Πολλά από τα σκάφη μας έχουν χαθεί και πολλοί αλλοίς ε, βασίζονται σε άλλα είδη. Με γαριδούλες, ψαρεύουν γαριδούλες. Σε ένα μικρό λιμανάκι πήγα στο Όμπι. Εδώ και δύο Σάββατα πήγα εκεί και το κουβέντιασα το θέμα με τους ψάραδες. Τα βρίσκουν σκούρα. Πολλοί μπορεί να φύγουν από τον τομέα πριν η μεταρρυθμίση δώσει αποτελέσματα. Υποχρεώθηκαν να ψαρεύουν γαρίδες, μικρές γαρίδες. και στην οικονομική κατάσταση και επειδή έχει κατακλειστεί η αγορά με γαριδούλες, ε, έχουν πέσει οι τιμές και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ένας νέος που έχει οικογένεια και τέσσερα παιδιά. Μου ήρθε μετά από τη συζήτηση Τετάρτη και είπε ότι έχασε 850 λίρες τερλίνες στην προσπάθεια που έκανε. Πολλοί θα συμφωνούν μαζί μου όταν λέω ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για πολλούς ψαράδες. Ψαράδες που ζουν σε μικρές κοινότητες, στις ακτές της Βορείου Ιρλανδίας. Άκουσα με ενδιαφέρον αυτά που υπόθεκαν. Και βέβαια τα δημόσια χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργούνται δουλειέ. Αλλά έχουμε καθήκον να δημιουργήσουμε και βιώσιμε κοινότητε. Και πολλέ από τι κοινότητε τη Βόρεια Ιρλανδία εξαρτώνται από το ψάρεμα. Για να επιβιώσουν. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πολλοί ψαράδες και εκπρόσωποι του τομέα που συναντάω θα ενθαρρυνθούν από κάποια από τα σχόλια που άκουσα σήμερα ο τομέας και εγώ θα καλωσορίζαμε περισσότερη συμμετοχή στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Να έχουν λόγο οι ψαράδες περισσότερο. Αισθάνονται σαν να τους επιβάλλονται λύσεις. Δεν τους ζητάμε να συνεργαστούν, να εκφράσουν άποψη. Και με ενεθάρρυναν αυτά που άκουσα. Θα πρέπει να το αναπτύξουμε αυτό και να συνεργαστούμε με προσώπους του τομέα όλες οι περιοχές να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Πολλοί εκπρόσωποι που συναντώ έχουν βαρεθεί με τη μικροδιαχείριση της περιφερειακής αλίας που γίνεται τις Βρυξέλλες. Θέλουν τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν λόγο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Αισθάνονται ότι αν είχαν αντιμετωπιστεί τίτο τρόπος θα μπορούσαν να δώσουν κάτι με αίσθημα ευθύνη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να τονιστεί. Εν κατακλείδη έχω να πω τρία πράγματα. Τα θεωρώ σημαντικά. Που ίσως αυτά τα τρία στοιχεία μπορούν να μας κατευθύνουν σαν Επιτροπή όταν εξετάζουμε τη μεταρρύθμιση. Ποια είναι αυτά. Σε αυτό το επίπεδο θέλουμε γενικές αρχές, κατευθυντήριες αρχές θα πρέπει η διαχείριση να φύγει από το κέντρο και να πάει στην περιφέρεια. Εκεί αυτοί οι ντόπιοι που ξέρουν την περιοχή και εργάζονται εκεί και ξέρουν πώς ζει η περιοχή από τον τομέα και πώς μπορούν να κάνουν τον τομέα βιώσιμο, αυτοί να μπορούν να έχουν λόγο. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στη διαδικασία. Θα υπάρχουν και δύσκολα ζητήματα αλλά τα δύσκολα θέματα θα είναι λιγότερα αν συμπεριληφθεί ο τομέας και οργανώσεις των αλλιέων στην διαβούλευση. Αυτή η Επιτροπή, και εγώ μιλάω σαν νέο μέλος της Επιτροπής και νέο μέλος του Κοινοβουλίου, αυτή η Επιτροπή λέγω ακολουθεί ένα δρόμο που ίσως οδηγήσει σε ένα ευπρόσδεκτο ταξίδι για την Ευρώπη. Μιλώ εγώ που θα ήμουν κατά της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης και θα πρέπει να δώσουμε πραγματική εξουσία στον κόσμο που ξέρει την περιοχή του, να ζητήσουμε από αυτούς να διαχειριστούν την περιοχή τους, να ζητήσουμε από αυτούς να ετοιμάσουν μακροπρόθεσμα σχέδια για μια μακροχρόνια βιώσιμη αλληλεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε το λόγο τώρα στον κύριο Γκρόμπατσικ. Συγγνώμη αν δεν, αν δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας, αλλά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Με χαρά. Ακούω αυτές τις προτάσεις και αυτά που συμπεριλαμβάνει η πράσινη βίβλος όσον αφορά την περιφερειοποίηση της πολιτικής, διότι αυτό είναι σημαντικό για τους αλίες. Πρέπει οι νόμοι να μην καλύπτουν όλους με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την τοπική κατάσταση. Το ανέφερα και στο παρελθόν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πολιτική να λάβει περιφερειακό χαρακτήρα. Και οι διατάξεις να θεσπίζονται συναρτήσει των τοπικών συνθήκων. Αυτό είναι σημαντικό. Στις περιοχές αυτές που χαρακτηρίζονται και από ιδιαιτερότητες. Είναι σημαντική συνεργασία με τους κύκλους των αλλιών πρέπει να ενεργοποιηθούν οι αλλιείς, να κινητοποιηθούν, ούτως τόσο να συμμετάσχουν στην ε, περιφερειοποίηση της πολιτικής. Κάτι που θα σημάνει ένα νέο άνοιγμα της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, διότι μέχρι τώρα αυτή η πολιτική δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το σημαντικότερο θέμα είναι το εξής. Αν θέλουμε να αλλάξουμε πολιτική, θα πρέπει να κάνουμε σωστές εκτιμήσεις των αλληλευτικών πόρων που υπάρχουν στις διάφορες ζώνες. Εδώ δημιουργείται η αντίθεση μεταξύ του κόσμου των αλλιών και του επιστημονικού κόσμου, διότι μεν και οι δε έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις. Και πρέπει αυτό να λυθεί. να βρούμε. Χρειάζεται μείωση ελευτική προσπάθεια. Δεν χρειάζεται. Πού χρειάζεται. Και αν πρέπει να καταλήψουν τον τομέα οι αλληλείς και να βρουν ένα άλλο επάγγελμα, να μπορούν να το κάνουν αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπενθυμίζω την κατάσταση της Βαλτικής, με τη Ρέγκα και άλλα είδη. Εδώ και δύο χρόνια έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μικρή αλληλείς θα έπρεπε να αλλιεύουν δύο συγκεκριμένα είδη. Ότι είναι μονο, θάλασσα μονοκαλλιέργειας. Ότι υπάρχει μόνο μπακαλιάρος στην Βαλτική. Η κατάσταση άλλαξε όμως έκτοτε. Υπάρχει μείωση φοβερή των ειδών αυτών και μειώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ποσοστώσης. Βλέπουμε συνέπεια πλήρης ασυνέπεια επικρατεί στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Τι θα γίνει λοιπόν. Άλλο ερώτημα. Σχέση μεταξύ οικονομίας και αλληλευτικού τομέα. Εδώ είναι προφανέστατο το συμπέρασμα. Όσον αφορά τους μικρούς αλληλείς, σε σχέση με τη βιομηχανική αλληλεία πάντα χάνουν αυτοί. Πάντα κερδίζει η βιομηχανική αλληλεία παράγουν αμέσως από την αλληλεία ηχθιάλευρα, οι μεγάλες εταιρείες, και πουλούν τα ηχθιάλευρα με έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου επωφελής για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω το πρώτο κατάλογο αυτούς που σημείωσα. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην εφημερίδα και μετά έχουμε στι 5.30 τους usted. Eh, señor Haglund, señor Hacton, señor André, Andrés Barea, señor Gallagher, señor Davis y señor Antinoro. Y con esto luego intervendrá la comisión si quiere la ponente y cierro la lista. Señor eh, Haglund. Κλείνει με αυτού η λίστα των αγορητών και πρώτο λαμβάνει το λόγο ο κ. Χάρτλοντ. Tack, bästa ordförande, kollegor. Eftersom tiden då tydligen håller på att ta slut så ska jag fatta mig kort och inte upprepa. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα είμαι Σύντομο, δεν χρειάζεται να επαναλάβω όσα υπόθηκαν πιο πριν. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ καλό που μπορώ να συνεχίσω από εκεί που τελείωσε ο προλαλή σα. Ε, πρέπει όντω να επικεντρωθούμε στους ε, μικρούς ε, αλληλεί. Η πράσινη βίβλος έχει μια τέτοια πτυχή. Βέβαια, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στην πράξη. Καλή είναι η θεωρία πρέπει να ορίσουμε ε, πώς είναι, ποια είναι η μικρού επίπεδου, μικρού εύρους αλληλεία, ποιο είναι, ποιο είναι το φάσμα το οποίο μετρούμε. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες οι προϋποθέσεις που θα θέσουμε ε, να τηρούνται βεβαίως οι καταστάσεις είναι διαφορετικές ανάλογα και με τη θάλασσα που αλλιεύει κανείς υπάρχουν ούτως ή άλλως τέτοιες ε, διαφορές πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί αναλόγως και ο ορισμός υπάρχουν ε, διαφορετικές ζώνες αλλιείας και η συνάδελφος από την Ιρλανδία μας είπε ότι όντως υπάρχουν προβλήματα η καθοδήγηση από, την, ε, από τις Βρυξέλλες πρέπει να φτάνει μέχρι ενός σημείου και θα πρέπει όντω οι αποφάσει που λαμβάνονται να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στην πρακτική, όσο δυνατόν πιο κοντά δηλαδή στις περιφέρειες. Προς τα εκεί πρέπει να, κινηθούμε, να κινηθούμε λοιπόν. Γιατί θεωρώ ότι έτσι μόνο θα λύσουμε το πρόβλημα και προς το παρόν έχουμε ξεκινήσει καλά, πιστεύω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τις αρχές που αναφέρθηκαν. Όντως, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ανάληψη της ευθύνης ε, και ε, αυτή η επικέντρωση όλων των ε, εξουσιών στις Βρυξέλλες είναι ένα κομμάτι του προβλήματος. Άκουσα την εισηγήτρια να αναφέρει διάφορους τομείς που πρέπει να επανεξεταστούν και τελείωσε με το ότι ναι πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση. Εγώ θα ήθελα να καλέσω την εισηγήτρια αυτή την αποκέντρωση και την περιφερειοποίηση να τη βάλει στις πρώτες θέσεις του καταλόγου για τις ε, άμεσες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσει από εκεί αντί να ξεκινάει από την ΚΑΠ όσα έχει. Όλοι τώρα δεχόμαστε ε, ότι η ΚΑΠ ήταν αποτυχημένη. Ε, θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο εάν προσεγγίζαμε το θέμα με τον τρόπο αυτό. Να δούμε δηλαδή ποιε είναι οι ε, διάφορε απόψει που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη διαχείριση συγκεκριμένων περιοχών, περιφερειών, για το ε, ποιο θα πρέπει τελικά να λαμβάνει αυτέ τι αποφάσει για του διάφορου τομεί κατά τη διάρκεια τη μεταρρύθμιση. Εγώ είμαι από τη Σκωτία και μα ενδιαφέρει φυσικά πάρα πολύ η Βόρεια Θάλασσα, για παράδειγμα. Ε, πρέπει λοιπόν τα πράγματα να είναι σαφή. Εμένα η δική μου εντύπωση είναι ξεκάθαρη. Τα τα αλληλευτικά μας δικαιώματα στην ε, Βόρεια Θάλασσα ε, θα πρέπει να μας δίνουν το δικαίωμα να έχουμε και λόγο στην οργάνωση των πραγμάτων για τη Βόρεια Θάλασσα. Ή τέλο πάντων ο καθένα ε, για την θάλασσα στην οποία αλλιεύει ή ενδιαφέρεται. Θα πρέπει λοιπόν οι ντόπιοι, οι άνθρωποι που λειτουργούν στα μέρη αυτά, να έχουν και λόγο. Έτσι ώστε να είναι και κατάλληλη η διαχείριση και τα μέτρα που θα λάβουμε στι ανάγκε τη συγκεκριμένη περιοχή. Απ' την άλλη, η ΚΑΠ έχει αντιμετωπίσει και άλλα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η έλλειψη πρωτοβουλειών για να συμμορφωθούμε με, τα... με τις ε, διαταγές, ας πούμε, που έρχονται άνωθεν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από πάνω προς τα κάτω για την διατήρηση των πόρων. Αν αλλάξει αυτό, θεωρώ ότι θα αποτελέσει ε, όθεση για την ε, ανάληψη πρωτοβουλειών για την ε, κάθε περιοχή. Προς το παρόν δημιουργούνται πάρα, πολλές, πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά το ποιο έχει την εξουσία για την, στα πλαίσια της παρούσας ΚΑΠ. Για τα τάκη της προσωστώσης τώρα. Αν προσεγγίσουμε τα πράγματα με τον τρόπο που θεωρώ εγώ, να γίνει δηλαδή αυτή η αποκέντρωση της λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να αποκεντρώσουμε και τα, τα των τάκτη ποσοστώσεων. Να γίνει ας πούμε μια κατανομή προσπάθειας. Ε, ο Επίτροπος όταν ήταν ε, εδώ, μας είπε ότι αυτά είναι εμπορεύσιμα δικαιώματα. Ε, αυτό εντάξει, εμένα μου ανάβει λίγο τα λαμπάκια, γιατί παραπονούμεθα από τη μια έντονα για τις ε, ε, δυνάμεις της αγοράς και το πώς δρούν σε ό,τι αφορά τους ε, λιανοπολιτές που μειώνουν τις τιμές. Απ' την άλλη πάλι φαίνεται ότι υπάρχει έτσι και κάποιο υποτιθέμενο όφελος ε, παραδίδοντας την, τα δικαιώματα αυτά σε αυτές τις δυνάμεις της αγοράς. Όντω μπορεί να υπάρξει οφέλο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε με μια κατάσταση η οποία να μην οδηγήσει σε ένα μικρό αριθμό πολυεθνικών οι οποίες θα έχουν αγοράσει όλα τα αλληλευτικά δικαιώματα. Εμένα δεν με νοιάζει το πού θα γίνονται αυτές οι δραστηριότητες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι αρκετό για μας να δεχτούμε ότι αν επί της αρχής συμφωνήσουμε ότι όντως θα υπάρχουν αυτά τα, ένα σύστημα με δικαιώματα και προσπάθεια, θα αφήσουμε στην Κομισιόν τα υπόλοιπα να ορίσει δηλαδή ποια είναι η ε, αλληλεία μικρής ε, κλίμακος. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει η συγγήτρια. Ότι δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε έτσι να οριστεί τι είναι η αλληλεία μικρής κλίμακας αντί να περιμένουμε από την Κομισιόν να αποφασίσει πρώτα επί της αρχής και μετά να μας υποβάλει μια γνωμοδότηση επ' αυτού. Γιατί η μικρή κλίμακα σε μια περιοχή μπορεί να σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό σε μια άλλη περιοχή. Και επανέρχομαι σε αυτό που, ε, από το οποίο ξεκίνησα. Γιατί δεν έχουμε μια πολιτική η οποία να δίνει τη δυνατότητα αυτές οι αποφάσεις να λαμβάνονται επιτόπου στις περιοχές που τις αφορούν από τους ανθρώπους που τους αφορούν. Και κλείνοντας, εδώ να πω ότι το πώς όλες αυτές οι αρχές μπορούν να μεταφραστούν σε ένα νέο σύστημα θα πρέπει όντω να αναφερθεί σαφώ. Ούτω ή άλλω οι, οι βασικέ αρχέ είχαν λόγο ύπαρξη όταν εκπονήθηκαν. Και τέλο, η ΚΑΠ που έχουμε τώρα λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση στα ύδατα και στους πόρους. Για τα ευρωπαϊκά πάντα μιλούμε. Και πάντα θα υπάρχει αυτή η απειλή, ας πούμε, που θα αφορά τις μεταρρυθμίσεις για οποιοδήποτε άλλο τομέα γίνουν. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Ο Επίτροπος είπε ότι δεν θα ξεχάσει τίποτα. Αυτό και όντω δεν θα πρέπει να το ξεχάσει. σε ε, Παρακαλώ να είστε σύντομοι, αλλιώ δεν προλαβαίνουμε. Κυρία Μπαρία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο συγητή πάρα πολύ καλά τα είπε και μακάρι να ήταν τα πράγματα βέβαια όπω είπε, δηλαδή να μπορούσαμε να πάμε πέρα από την περιφερειοποίηση και να μπορέσουμε να σώσουμε και τη θάλασσα και τα λιμάνια και την αλληλεία και την απασχόληση. Άρα να γίνει μια προσπάθεια παραπάνω. Να ξανοιχτούμε λίγο παραπάνω δηλαδή στο πέλαγος μεταφορικά. Θα πρέπει να είναι το μήνυμα ξεκάθαρο τόσο ώστε να είναι κατανοητό για όλους τους συμπλεκόμενους, τους διαφορετικούς συμπλεκόμενους γιατί πρόκειται για διαφορετικά κομμάτια του κλάδου, διαφορετικών περιφερειών, διαφορετικών ε, συνηθιών ψαρέματος και έτσι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο σωστά τα δημόσια χρήματα και να είναι δυνατόν ο κλάδος να χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα την υπεύθυνη αλία, ε, ε, τα απορριπτώμενα ψάρια, τα τάκ. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι το να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με την αιτία στις τρίτες χώρες. Και συζητάμε τώρα για τις διεθνείς αλληλευτικές συμφωνίες που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει καμιά πόρτα, δεν, υπάρχει, δεν γνωρίζουν κανένα περιορισμό οι θάλασσες και το νερό. Οπότε και γι' αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια όσον αφορά τις ενέργειες υποστήριξης της Αγγλίας. Κύριος Αντιπρόεδρος, μα είπε ποια είναι τα νομικά προβλήματα και δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε εάν δεν προσυπογράψουν οι εμπλεκόμενες χώρες όλες τις σχετικές συμφωνίες και πάντοτε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν προβλέπονται κάποιε κυρώσει σε κάθε συμφωνία. Και αυτό βέβαια είναι αντικείμενο συνενετική αντιμετώπιση από όλε τι χώρε. Να κάνουμε επομένω μια τέτοια αξιολόγηση ευρύτερη παραπέρα από την περιφερειοποίηση και έτσι να καταφέρουμε να σώσουμε τη θάλασσα και την αλία αλλά και την απασχόληση. Τι ωραία τα είπε ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί στον τομέα που είναι αρκετά διστακτική όσον αφορά αυτήν την αναθεώρηση. Είναι κατανοητό, κατά παρελθόν είχαν γίνει ενδιάμεσα αναθεωρήσεις και δεν είχαν γίνει σημαντικές επίσης. Έγινε μια αλλαγή την περασμένη φορά και ήταν η δημιουργία των ΡΑΚΣ, των Περιφερειακών Συμβουλίων. Ήταν μια σημαντική εξέλιξη αυτή και σε αυτή την αναθεώρηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις που θα μας πούν οι υπεύθυνοι του τομέα. Γιατί το λέω αυτό. Διότι βλέποντας το μέλλον του τομέα, εάν δεν έχουμε μια αλληλεία, ποιος θα χάσει τα περισσότερα δεν είναι ο βουλευτή, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι το Συμβούλιο, αλλά ο τομέα. Και ενώ υπάρχει άποψη ότι ο τομέα θα είναι ικανοποιημένο όταν θα έχουν βγάλει όλα τα ψάρια τη θάλασσα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Θα δώσω ένα παράδειγμα, την προηγούμενη φορά όταν ήμουν εδώ. Όσον αφορά τα μέτρα τεχνική συντήρηση, ήταν μη προσέγγισε το κάτω προ τα άνω. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προερχόταν κυρίω από τη χώρα μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπήρχε υποστήριξη πολύ μεγάλη από τις άλλες χώρες, διότι τα τεχνικά μέτρα συντήρηση είναι πάρα πολύ σημαντικά, μέγεθος δικτύων, ούτω ώστε να μειώσουμε την ποσότητα των ε, απορρίψεων. Αυτοί έχουν περισσότερα πράγματα να χάσουν οι αλλοί, άρα είναι ζωτική σημασία αυτοί οι άνθρωποι να έχουν συμμετοχή στις συζητήσεις και ξέρω ότι θα υπάρξει αυτό και ξέρω ότι και η παραγωγή και οι μεταποιητές ε, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους σχετικά με το θέμα αυτό. Αυτοί έχουν τα περισσότερα να χάσουν. Τώρα τα τάκτη ποσοστώσεις ε, έχουν ενθαρρυνθεί. Έχουν γίνει διάφορες ε, δηλώσεις από τον Επίτροπο Μπόργκ, τον Επίτροπο και τελευταία φορά που συναντήθηκε είπε ότι θα το εξετάσουμε. Δεν τα είπε ο ίδιος, αλλά όλα είναι επιτάπητος είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος, εννοεί αυτά που λέει και δεν ε, λέει απλώς κάποια πράγματα. Όσον αφορά τα τάκ και τις ποσοστώσεις, είδαμε ότι δεν έχουν εξυπηρετήσει αυτά τα μέτρα εξής όλες τις χώρες, αλλά παρομοίως θα πρέπει να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε και αυτό, καθώς και τις μεταφερόμενες εμπορεύσιμες ποσοστώσεις. Βεβαίως, τα τάξ και οι ποσοστώσεις δεν βοήθησαν τις μικρές χώρες, οι οποίες δεν είχαν ισχυρό ιστορικό παρελθόν. Ίσως όσον αφορά τον αριθμό των μικρών σκαφών, όσον αφορά τις εκφορτώσεις ποσός, ε, όγκων, ε, οι χώρες όπως η δική μου έπρεπε να μοιράζονται ψάρια με άλλους που έμπαιναν στον τομέα. Γίνεται δημοψήφισμα την Παρασκευή στην Ιρλανδία και ελπίζω και όλα τα κόμματα θα περάσουν την συνθήκη. Αλλά ο τομέα είναι αυτό που έχει πέσει του λόγου να είναι αντιευρωπαίο. Διότι έχουν πληρώσει πάρα πολύ υψηλό τίμημα. Αλλά για να δείξουν ρεαλισμό και πραγματισμό, δύο από τι μεγάλε αλληλευτικέ οργανώσει. και οργανώσει παραγωγών Ιρλανδών υποστήριξαν το ναι. Και του συγχαίρω γι' αυτό, διότι καταλαβαίνουν ότι ένας τρόπος που μπορούμε να βελτιώσουμε τη μοίρα μας είναι εντός της κοινότητας να παίζουμε στο κέντρο του γηπέδου και όχι έξω από τις γραμμές και έτσι όλοι μας μπορούμε να έχουμε περισσότερη εξουσία και περισσότερη συμμετοχή στη συναπόφαση στο Κοινοβούλιο. Η αναθεώρηση ελπίζω ότι θα ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Σίγουρα όμως δεν θέλω ένα σύστημα το οποίο θα καταλήξει στο εξή. Άλλοι που μπορούν να αγοράσουν τις εμπορεύσιμες ποσοστώσει ή τα σκάφη να το κάνουν. Και μπορεί να χρησιμοποιούνται και σημαίε ευκαιρίες που έρχονται σκάφη και βάζουν Ιρλανδική σημαία για άλλου λόγους. Συγχαίρω την εισηγήτρια, μας έδωσε μια γενική εικόνα, αλλά πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειε και ελπίζω ότι οι απόψει που εκφράζουμε θα ληφθούν όντω υπόψη. Συμφωνώ με το συνάδελφο τη Βορείου Ιρλανδία Είναι πολύ σημαντική η περιφερειοποίηση. Η περιφερειοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ δεν έχουμε ένα γάντι που ταιριάζει όλα τα χέρια. Ένα και μόνο μέτρο χρειάζεται η άποψη του τομέα. Άλλο γίνεται στη Βόρεια Θάλασσα, άλλη κατάσταση στη Μεσόγειο, άλλη στη κατάσταση στη Βόρεια Θάλασσα, στη δική ακτή της Σκοτίας ή της Ιρλανδίας. Χρειάζεται περιφερειακό χαρακτήρα η προσπάθεια, περιφερειοποίηση χρειάζεται. Καλωσορίζω την ε, εφαρμογή των RACs. Πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε στα σοβαρά στην έκθεσή μας ένα κομμάτι που θα καλύπτει τα μικρά σκάφη. Κάποιο θα πει εντάξει ότι είναι κάτω από 10 μέτρα. Ναι βέβαια ότι είναι κάτω από 10 μέτρα. Αυτοί που είναι γενναίοι και ανοίγονται αυτά τα σκάφη και υπάρχουν ακτέ όπου υπάρχουν διάφορα ψάρια όπω μπακαλιάρο και ταξιδεύουν 7 ώρε αυτοί οι άνθρωποι. Βοηθήστε ε, να εξασφαλίζουμε την υγεία και ασφάλειά του. Πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα. 15 με 20 μέτρα. που έχουν ε, πολύ μικρή επίπτωση γενικά. Η επίπτωση της αλίας στα αποθέματα είναι αμεληταία. Αυτό πρέπει να εξεταστεί επίσης. Εν κατακλείδη, όποιοι από εμά έχουμε νησιά στην εκλογική μας περιφέρεια, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική απασχόληση για τους ανθρώπους στα περισσότερα μικρά νησιά. Καμία εναλλακτική. Λίγο τουρισμός, αλλά δεν είναι κάτι βιώσιμο αλλά υπάρχει η δυνατότητα με μικρά σκάφη που αλλιεύουν στα νησιά να μην πάνε σε άλλες χώρες, να επιστρέφουν στα λιμανάκια τους και να γίνεται και κάποια μεταποίηση εκεί. Λοιπόν, εισηγήτρια, μικρά σκάφη, ένα σημείο. Πόσα μέτρα το αποφασίζουμε. Και τα νησιά. Τι έγινε πρόσφατα. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν ε, κάποια είδη, πρέπει να επικεντρωθούν σε άλλα είδη να αλλάξουν, να πάνε στο στρακοειδή, να πάνε να ψαρεύουν ε, ε καβούρια, αστακού κλπ. Σταματήστε κύριε Γκάλα και σας παρακαλώ λέει πρόεδρο. Αν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ολοκληρώστε. Διότι δεν ε, μας μένει χρόνο, Να μην ξαρίσουμε το χρόνο με αυτό το θέμα. Τελειώστε παρακαλώ. Περιμένετε λέει ο κ. και συνεχίζει. Γιατί να με κόψετε εμένα κύριε πρόεδρε, λέει απτόητος ο κ. Γκάλακερ. Και αν εγώ γουστάρω θα συνεχίσω. Και θα πρέπει να έχω υπόψη το έτοιμά σα και όχι να μου το επιβάλλετε. Εκπροσωπώ το λαό μου. Και δεν μου αρέσει ότι εγώ υποχρεώνομαι να συντομεύω. Ίσως να είμαστε μικρότεροι, αλλά θα εισακουστούμε. Και ξέρω ότι η συγγήτρια θα λάβει υπόψη τις απόψεις μας, αν εσείς δεν τις λάβετε. yo tampoco voy a intervenir porque se ha acabado el tiempo. Yo soy la que cedo el tiempo a todo el mundo. Όχι, όχι. Όταν χρειάζεται, όταν ε, τελειώνει ο κόσμος, εγώ κόβω όποιον χρειάζεται. Δεν θέλω να ανοίξω διάλογο με σας κύριε Γκάλεχερ. Ντέιβις. Well, thanks, Chairman. Uh, may have been the first. I expect I'll be the second. Um... Ήταν ο πρώτος, ο κύριος Γκάλεχερ. Εγώ θα είμαι δεύτερος που θα κόψετε. Διότι πρώτα-πρώτα πήγαινε σε αποκέντρωση και για κεντρική διαχείριση. Δεν είμαι κατά. Παρά τότε η κατάσταση δεν είναι και τέλεια. Πάντως η Αλία δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τη συνθήκη όσον αφορά την κατανάθεση αρμοδιότητα, την αποκέντρωση και ελπίζω η Κομισιόν να είναι πιο αποφασιστική. Να έχει καταλήξει κάποτε να κάνει κοινέ προτάσει. Δηλαδή, ε, ε, σύμφωνα με τη συνθήκη, μέχρι πού φτάνουμε. Αλλιώ δεν συνοδεύονται από έργα τα λόγια μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Κάτι άλλο τώρα. Η κατάσταση αυτή είναι παράλογη, πρόκειται για έναν ε, φαύλο κύκλο, λιγότερη ελεία, λιγότερη θέση πασχόλης, λιγότερα χρήματα και κατόπιν μιλάμε για βιωσιμότητα. Να μπορέσουμε να έχουμε θάλασσες που αντέχουν περισσότερα ε, ψάρια ούτω ώστε να έχουν περισσότερο ψάρεμα, περισσότερες δουλειέ, περισσότερα λεφτά, ε, λιγότερες ε, εισαγωγέ που μας ρουφάει το κεφάλαιο. Πώς θα γίνει όμως αυτό, πώς θα αντιστρέψουμε αυτή την διαδικασία. Αυτό θα είναι επώδυνο. Και έτσι να μπορέσουμε να δώσουμε δουλειά στου ψαράτες, έστω και για λίγο. Και έτσι με κάποιο είδου διακοπή, αναστολή, τέλο πάντων οι ελευθερικοί πόροι να ανανεωθούν. Επομένω, παρακαλώ, η Κομισιόν, δώστε μα πολιτικό μήνυμα, δώστε καινούργιε προτάσει, ότι είναι δυνατόν να υπέρθει μια βελτίωση, αλλά αυτό θα γίνει με τρόπο επώδυνο, αν την ώρα. Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Διότι, όπως υπόθηκε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Η περιφερειοποίηση, η λέξη αυτή είναι το βασικό στοιχείο. Και στο τέλος συμφωνούμε όλοι πάνω σε αυτό, πιστεύω. Αυτή η μεταρρύθμιση ταυτόχρονα είναι και ελπίδα και σε κάποιες περιπτώσεις και μια απογοήτευση. Για αυτά που υπόθηκαν. Αυτοί είναι οι λόγοι που αναφέρθηκαν από άλλους. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες περίμεναν περισσότερα και απογοητεύτηκαν. Άρα δεν είναι απλός ο στόχος μας και το έργο μας. Περιγράφηκαν πράγματα από την εισηγήτρια και έχω μόνο κάτι να προσθέσω για να μην μακρηγορώ. Είναι δυνατόν. διαιρωτώ με απευθυνόμως με πρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την εισηγήτρια, από τις υπηρεσίε και κυρίως το, θέμα, το ερώτημα το απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχουν όρια στη θάλασσα, πράγματι υπάρχουν σύνορα. Στη Μεσόγειο όμω έχουμε περισσότερα προβλήματα από ό,τι υπάρχουν σε άλλα μέρη. Ε, ανέφεραν τι δικέ περιοχέ άλλοι συνάδελφοι. Στη Βόρεια Θάλασσα, μόνο οι λύσει τη Βόρεια Θάλασσα πάνε να ψαρέψουν και γυρίζουν στα λιμάνια για να επεξεργαστούν τα εναλία του. Στη Μεσόγειο δεν γίνεται αυτό. Έχουμε χώρες απέναντί μας που έρχονται σε εμά να ψαρέψουν δεν τηρούν τους κανόνες τους κοινοτικού, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι και υπάρχει ανισορροπία σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης. Τεράστια ανισορροπία, πολύ πιο μεγάλη από αυτή που διαπιστώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές θάλασσες. Και το ζουν αυτό οι πολίτες της Νότιας Ευρώπης και κυρίως της Νότιας Ιταλίας το αντιλαμβάνονται για άλλο, σαν άλλο ένα πρόβλημα, πέρα από τα προβλήματα λήψης απόφασης. Επισήμως ρωτώ και ζητώ αν μπορούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ίσως με τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεργαστούμε για να δούμε ότι εφόσον θα εξετάσουμε την πράσινη βίβλο που δεν αναφέρεται μόνο στην αλληλεία αλλά αναφέρεται και θα πρέπει να αναφέρεται και στα προβλήματα άλλα όπως σύγκρουση περι, ε, περιφερειακών αρμοδιοτήτων. Πού μπορεί να πάει κανείς, πού να αλλιεύσει, τι να αλλιεύσει. Διότι πιθανότατα η πράσινη βίβλος που θα είναι, και θα είναι λευκή βίβλος αργότερα θα αντιμετωπίσει το θέμα από μια γωνία και θα θεσπίσει μια αλλιευτική πολιτική που θα ξεπερνά τα όρια της ε, αλίας απλής αλλά και τις σχέσεις με άλλες χώρες. Είναι υποχρέωσή μου για μένα που ζω αυτά τα προβλήματα και προσωπώ αυτή την περιοχή της Ευρώπης να εκφράσω αυτά τα προβλήματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν θα λάβω το λόγο. Για να μην εκνευριστεί κανείς, θα πάρει την πρώτη λόγο η ε, Επιτροπή. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί βλέπω ότι έχει πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να απαντήσω σε όλους μαζί, αν γίνεται, για τρία-τέσσερα σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι αυτά που αποτελούν την ουσία αυτής της μεταρρύθμισης. από τα πρώτα σε σχέση με τους Ιρλανδούς αλλιείς, που είναι οι πρώτοι που αντιτίθενται σε αυτή την πολιτική. Προσοχή διότι 20 χρόνια που δουλεύω στην Ελία αναπτύχθηκαν οι Ιρλανδοί σε αφορά την Ελία λόγω της Ευρώπης, λόγω της Ένωσης. Και μέσα οι επιβαρύνσεις αναλογικά βαρύνουν όλους. Να μην ξεχνούμε επομένως ότι κατά τη γνώμη μου ωφελήθηκε πολύ από την ΚΑΠ Ιρλανδία. Αυτό είναι γεγονός, πραγματικό περιστατικό, δεν είναι πολιτική αξιολόγηση. Τα δικαιώματα της Ελίας είναι εξατομικευμένα, είναι μεταβιβάσιμα και είναι κάτι το οποίο αφορά αυτή την προσπάθεια μεταρρύθμισης γιατί θέλουμε να δούμε ποια είναι η κλίδα κατανομής των σχετικών δικαιωμάτων κάτι πρέπει να είναι σύνομο με το κοινοτικό δίκαιο, με το δίκαιο της σημαίας και τις διατάξεις που διέπουν την ΚΑΠ. Να ποια είναι η ουσία αυτή της μεταρρύθμισης. Η καρδιά τη μεταρρύθμισης, κάτι άλλο το οποίο εδώ τονίσατε που είναι σημαντικό και έχετε δίκαιο, είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπορκ, ο Επίτροπος Ελίας, ότι δηλαδή θα πρέπει τα ΤΑΚ να υποστούν κάποια μεταρρύθμιση. Αυτό είναι απαραίτητο, έχει προκύψει σε πολλές περιπτώσεις, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη μεικτή αλία. Υπάρχουν όμω κάποιε τεχνικέ δυσκολίε και χρειάζεται κάποια μεταβατική περίοδο όσον αφορά τη μεταβασία από το ένα σύστημα στο άλλο χωρί να μην υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση σε κανέναν. Χρειάζεται κάποια προσαρμογή και αυτό είναι θέμα που χρειάζεται εξέταση, που και αυτό είναι σημαντικό στη μεταρρύθμιση. Άλλο, σωστά το επισημάνατε, είναι η περιφερειοποίηση. μικροδιαχείριση, περιφερειοποίηση, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες, να μπορούμε να δώσουμε επίσης περισσότερες εξουσίες στους αλληλείς, στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Σε σχέση με, τα, με το συμφέρον της κάθε περιφέρειας και του οικοσυστήματος. Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν πολιτικά θέματα, θέματα κοινωτικού δικαίου. Γιατί είναι δυνατόν να ανατεθούν αρμοδιότητες περισσότερες σε κάποιους ε, φορείς. Και αυτό το προβλέπει η μεταρρύθμιση. Επίσης, αυτή την παράκτη αλληλεία για μας είναι κάτι το οποίο είναι αλληλένδετα συνδεδεμένο με το πώς θα διαμορφωθούν τα δικαιώματα αλληλείας την επαύριο και πώς θα γίνει η εξατομίκευση και τι είδους μεταβιβασιμότητα θα υπάρχει προστασία του αλλιεύματος θα πρέπει να διέπεται και στην περίπτωση της υπαραγωγής αλλιείας από τις ίδιες αρχές όπως κάθε είδους αλλιεία. Απομένως, η βιωσιμότητα των πόρων ακριβώς όπως ε, ισχύει και για τις, τα υπόλοιπα είδη αλλιείας. Είναι κάτι επομένως το οποίο έχει σχέση με την κοινωνική διάσταση της ΚΑΠΑ έχει σχέση και με την επιμέλεια του περιβάλλοντος και είναι θέμα αυτής της μεταρρύθμισης. Και Πρόεδρος, κύριε Πατρά, έχει το λόγο για να ολοκληρώσω. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα όλες τις ε, απόψεις Βέβαια είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε και αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ είναι να αναφέρω ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και επί τη βάση συνένεσης ε, να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Προσπάθησα επίσης να σκιαγραφίσω ε, πού είναι, ποιοι είναι οι φορείς, που, οι τομείς μάλλον που πρέπει να δράσουμε και να δούμε πού μπορούμε να ε, κάνουμε την ε, διαφορά. Βέβαια πολλά έχουν να κάνουν και με το πώς διαβάζει κανείς την πράσινη βίβλο και πώς θέλει να φτάσει στη λύση που χρειάζεται. Πολλά λοιπόν θα εξαρτηθούν από την οπτική γωνία του καθενός και από το πού θα αποφασίσουμε ότι θέλουμε να φτάσουμε τελικά. Φυσικά θα υπάρξουν και κάποιοι τομεί για του οποίου θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, περιφερειοποίηση όπως ακούστηκε πιο πριν, επίσης η συμπερίληψη όλων, όλων των φορέων που εμπλέκονται σε δραστηριότητε αλληλεία. Και αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να εξευρεθεί ο μέγας συμβιβασμός. Υπάρχουν φυσικά και συγκεκριμένα προβλήματα και φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνήσουμε επ' αυτού. Το θέμα δεν είναι να βρούμε μια λύση που να κάνει σε όλους, ε, δεν είναι πανάκια. Ε, πρέπει να καλύψουμε όχι μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε και κάποιες βασικές προϋποθέσεις για, στα πλαίσια ενός συμβασμού. Κάποιοι θα πρέπει να κάνουν ε, θυσίες. όντως θα χρειαστεί να υπάρξει συμβιβασμός από κάποιους. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε, να διαγράψουμε, να λύσουμε μάλλον προβλήματα του παρελθόντος. Να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς που πλήττονται ιδιαίτερα. Έγιναν και κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τις ιδέες που μου δώσατε. Αν έχετε και άλλες ανησυχίες, πείτε μου. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να έχω υπόψη μου, πείτε μου, πείτε μου το, για να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσουμε με αυτή τη ε, συζήτηση, ούτως ή άλλως και το Νοέμβρη. Πάμε τώρα στο σημείο 8 Λυπάμαι που έχουμε λιγότερο χρόνο από έχουμε αρχικά ε, προβλέψει, κύριε Μιλάνα. Πρόθεση τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη τη ευρωπαϊκή αυτοκαλλιέργεια. Ο κύριο Μιλάνα, ο συγκητή, θα του δώσω αμέσω το λόγο. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε, να είμαι εξαιρετικά σύντομο. Και επειδή εδώ είμαστε στην ε, φάση που ο εισηγητής θα πρέπει μάλλον να ακούει παρά να εκθέτει την ε, δική του άποψη. Η ανακοίνωση της Κομισιόν έρχεται πολύ, χρονική, πολύ καλή χρονική στιγμή. Είναι γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη από το 2002 και έχουμε φτάσει σε μια πολύ ευαίσθητη ε, κατάσταση για τον κλάδο. το οικονομικό μας πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό. Ζητά πραγματικά πολλά για τα για την υδατοκαλλιέργεια, όχι μόνο για την ε, Ευρώπη. Πρέπει να δούμε και την ε, ανάπτυξη που έχει υπάρξει, η οποία ήταν στις τάξεις του 6 με 8%. Εμείς έχουμε αναπτυχθεί πραγματικά πολύ λιγότερο από όλο τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Η περισσότερη ε, ανάπτυξη έχει υπάρξει στην Ασία και την Νότια Αμερική. Μιλούμε δηλαδή για ένα κύκλο εργασιών 3 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ σε άλλες ε, χώρες. Τώρα εμείς έχουμε σημαντικό πρόβλημα και με τις ε, εισαγωγές Υπάρχει μεγάλη ζήτηση περίπου για 12 δισεκατομμύρια τόνους μιλούμε εισαγωγών, που είναι πραγματικά ε, σημαντικό κομμάτι της γενικής ε, ε, ποσότητας. Η δική μας λοιπόν η δατοκαλλιέργεια είναι πολύ σημαντική να αναπτυχθεί. Μπορεί το δικό μας προϊόν να είναι καλύτερο, αλλά πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί ταυτόχρονα. Αν δείτε την ανακοίνωση 2011 και το 2002, θα δείτε ότι ε, αυτό που παράγουμε εμείς είναι ανεπαρκές. Και μάλλον και εμείς είμαστε τελικά ανεπαρκείς. Η σημερινή ανακοίνωση που είναι μεν καλή και πραγματικά καταδεικνύει ποια είναι η κατάσταση. Ε, βέβαια η βίβλο αυτή δεν είναι ούτε πράσινη ούτε άσπρη, είναι γκρι. Έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά και κάποια άλλα τα οποία χρήζουν επεξεργασίας. Η Γενική Διεύθυνση Αλίας υποβάλλει την, την ανακοίνωση αυτή. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, εγκρίνει τον ε, κανονισμό, το σχετικό κανονισμό. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την ε, βιοπαραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι σημαντικός ο κανονισμός, είναι πολύ περίπλοκος. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της βιολογικής καλλιέργειας. Βεβαίως θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν γίνει διαφορετικά, γιατί Όντως η καλλιέργεια είναι ένας τομέας ο οποίος έχει το δικό του ειδικό βάρος. Πρέπει όμως να ξεπεράσουμε και αυτό. Η ανακοίνωση από τον Απρίλιο του τρέχοντος δεν, δεν κάνει καμία αναφορά στον κανονισμό που εγκρίθηκε. Βέβαια είχαμε θετικά αποτελέσματα από τις ε, πολιτικές που έχουμε ακολουθήσει. Είχαμε ε, Είχαμε θετικά αποτελέσματα από τις πολιτικές που ακολουθήσαμε. Βεβαίως δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε πλήρως την συνολική ζήτηση. έχουμε μικρές ε, μονάδες υδατοκαλλιέργειας, αλλά έχουμε και μεγάλες μονάδες, ε, βιομηχανικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Και όντως αυτές είναι διαφορετικές. Κάποιες από τις μικρές ε, μονάδες έχουν γίνει μεγάλες τελικά. Και μάλιστα είμαι σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τεχνικό, τεχνολογικό επίπεδο, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις είναι και καρπός και αποτέλεσμα επενδύσεων όσον αφορά την έρευνα. Υπενθυμίζω και θα είμαι συνοπτικός γιατί πηδάω από θέμα σε θέμα αλλά υπενθυμίζω ότι το 98 εκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο δόθηκαν για καινοτομία και έρευνα στον τομέα. Τα ο... Ε, αυτά τα χρόνια πρέπει να δοθεί χώρος για άδειε. Η συμπεριφορά στην Ευρώπη ήταν σχιζοφρενική όσον αφορά τη χορήγηση αδειών και ήταν αυστηρέ οι προδιαγραφέ και διατάξει, διότι υπάρχουν όσον αφορά τη βιωσιμότητα αυστηρέ διατάξει και ποτέ δεν μετετράπησαν σε αξιοποίηση οικονομική. Προστιθέμενη αξία αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια ερμηνεία που δίνω στην όλη ανάγνωση του θέματος, δηλαδή η δυνατότητά μα που υπάρχει να έχουμε υδατοκαλλιέργεια βιώσιμη δεν μεταφράζεται σε προστιθέμενη αξία οικονομική. Οι δεσμεύσει είναι πολύ μεγάλες, αλλά δεν από αυτά, αυτές οι άκαπτες διατάξεις δεν είχα μεγάλο κέρδος. Πρέπει οι δεσμεύσεις και τα όρια να γίνουν ε, κάτι πιο σταθερό, αλλά η προστιθέμενη αξία να είναι καλύτερη, να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Δηλαδή, να βρούμε τη σωστή απάντηση όσον αφορά τι καλλιέργειες και τις εταιρείε που κινούνται σε τομέα. Θα οριμάσουν τα πράγματα την παράδοδο του χρόνου δεν, θα έχουμε, δεν χρειάζονται γενικές πολιτικές που κάναμε μέχρι τώρα, ούτε ανακοινώσεις εξ αποστάσεως, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε διατάξεις πιο οργανικές. Δεν ξέρω, μπορούμε να βρούμε έναν κανονισμό, μια οδηγία. Αυτή είναι η απάντηση. Αλλά πιστεύω ότι ο τομέα είναι αρκετά όριμο να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν εντό τη μεταρρυθμίσεω τη κοινή αληθική πολιτική ή παράλληλα μπορεί να γίνει μια πιο συνεκτική νομοθεσία. Προσωπικά, και το λέω αυτό με το μέγιστο δυνατό βαθμό ανοίγματο, ε, θεωρώ ότι καλύτερο θα ήταν κανονισμό. Κανονισμό που θα λαμβάνει υπόψη τη μεταρρύθμιση τη κοινή αληθική πολιτική, αλλά που θα είναι κάπω όπω έχουμε κανονισμού που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα τομεακή εντό τη κοινή αλληλευτική πολιτική Φερρυπίν. Ο κανονισμός θα πρέπει να συνοψίζει τις προτάσεις πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες. Σήμερα δεν υπάρχει γενική, γενικό πλαίσιο. Σήμερα έχουμε μεθοδολογία για την ε, ανατροφή των ειδών, ε, πώς χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα, τα φάρμακα, ε, τα πώς κατασκευάζεται μια εγκατάσταση, τι χαρακτηριστικά τεχνικά πετούνται ε, και είναι εκτός πλαισίου. Θα πρέπει λοιπόν να ετοιμάσουμε μια γενική, γενικό πλαίσιο καλλιέργειες, κάνοντας διάκριση των τριών τομέων. Ε, έχουμε τα, τα ψάρια του γλυκού νερού ε, και έχουμε και τις άλλες καλλιέργειες που είναι διαφορετικές. Η βιωσιμότητα των τριών ειδών υδατοκαλλιεργιών, ε, είναι διαφορετική. Ο τρόπο κατασκευή των εγκαταστάσεων είναι διαφορετικό, οι συνέπειε για το περιβάλλον είναι διαφορετικέ, άρα χρειάζεται μία εμβάθυνση. Συνοπτικέ κρίσει ακούστηκαν για τον αρνητικό χαρακτήρα τη υδατοκαλλιέργεια, αρνητικέ συνέπειε, που μπορεί να προέρχονται και από άλλε καλλιέργειε. Αυτή η κρίση όμω ε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε συγκεκριμένο είδο υδατοκαλλιέργειε ψάρια, ψάρια του γλυκού νερού ή άλλη ιδετοκαλλιέργεια. Πρέπει να έχουμε αυτού του τρει βασικού πυλώνες για την ιδετοκαλλιέργεια, εφαρμόζοντα την επικουρικότητα. Και οι τοπικοί φορεί να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Να πω δύο πράγματα. Σκεφτείτε τα. Χρειάζεται διαδικασία τυποποίησεως ε, των διαφόρων διαδικασιών υδατοκαλλιέργειας σε κάθε κράτος. Μπορεί να ακολουθηθεί μια προσέγγιση για να τυποποιηθούν οι πρακτικές και για την εγκατάσταση των ε, υδατοκαλλιεργιών και για τα συστήματα που θα ισχύουν για το μεγάλωμα των ε, ψαριών. Χρειάζεται βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και πρέπει να τα κάνουμε αυτά για να είναι βιώσιμοι. Και ο τίτλο ανακοινώσεώ μου είναι ακριβώ αυτό η βιωσιμότητα των υδατοκαλλιεργιών. Θα πρέπει να δούμε το ρυθμιστικό χαρακτήρα των παρεμβάσεων. Να βγούμε από την αστική προσε... να βρούμε ένα είδος αστικής προσεγγίσεως για τη θάλασσα, αν θέλετε, ένα σχέδιο ρυθμιστικό των παρεμβάσεων. Πού βρίσκονται οι καταστάσεις. Συναρτήσει των περιφερειών σχέδια που θα εγκρίνονται με λεπτομέρεια. Υδατοκαλλιέργειες και τουρισμός. Τι σχέση υπάρχει. Υδατοκαλλιέργεια προστατευμένες περιοχές. Υδατοκαλλιέργειες περιβαλλοντική κίνδυνη σημαντική. Λοιπόν, ένα, μια τέτοια προσέγγιση οργανωτική όσον αφορά τις θάλασσες είναι βασικό στοιχείο που πρέπει να ακολουθηθεί σχεδιασμός χρειάζεται όσον αφορά τις εγκαταστάσεις εδωκαλλιεργιών. Χρειάζεται και απλούστευση διοικητική. Συνοπτικά θα αναφερθώ, αλλιώ θα μονοπολίσω το λόγο, θα μιλάω μόνο εγώ. Ο κανονισμός προβλέπει ειδικό ταμείο που θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ενισχύεται η έρευνα και οι προδιαγραφές για την έρευνα θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο έρευνα, νέες τεχνολογίες, κατάρτιση. Τρία θέματα σημαντικά. Χωρίς αυτά, αυτές οι εγκαταστάσει ποτέ δεν θα είναι βιώσιμε. Υπάρχει αρνητική συνέπεια σε κάποιες εγκαταστάσει λόγω καταλήπων που δημιουργούνται από αυτέ τι εγκαταστάσει που μέσω προθυμένες τεχνολογίας που μπορεί να εφαρμοστεί μπορεί να μειωθούν οι αρνητικέ συνέπειε στο περιβάλλον από τα απόβλητα αυτών των εγκαταστάσεων. Η έρευνα ε, μπορεί να τονωθεί μέσω επενδύσεων. Κατάρτιση. Και αυτό μπορεί να καλυφθεί από τον κανονισμό. Μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών εν γέννη που συνδέονται με αυτού του παράγοντε χρειάζονται και άλλα θέματα σημαντικά δύο. Η ανταγωνιστικότητα και η αγορά. Είναι σαφέ ότι η ανταγωνιστικότητα όσο μα αφορά επιτυγχάνεται όχι μόνο όχι μέσω της μειώσεως των δαπανών, μείωση του κόστους. Διαφορετική προσέγγιση από ό,τι ακολουθούν στην Ασία και στην Νότια Αμερική που είναι βασικοί μα ανταγωνιστέ ή κάποιε μεσογειακέ χώρε που ασχολούνται τώρα, αρχίζουν να ασχολούνται με την καλλιέργεια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε τι δραστηριότητέ μα επί τη ποιότητα. Η ποιότητα δεν είναι κάτι αυτονόητο. Δεν αρκεί να πούμε ότι έχουμε ένα καλύτερο ποιοτικά προϊόν, η ποιότητα είναι αποτέλεσμα δράσεων. Χρειάζεται λοιπόν στον κανονισμό και στο γενικό πλαίσιο για αυτές τις θετικολιέργειες να προβλέπεται η βελτίωση της διατροφής των ζώων, να υπάρχει ανιχνευσιμότητα των ψαριών. Λόγω χρονικού δεν επισέλθω σε λεπτομέρειες, βελτίωση της διατροφής πρέπει να συνοδεύονται και από ένα σήμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν περιθώρια και είναι σημαντικότατο τομέα. Εκτό η βιολογική υδατοκαλλιέργεια μπορεί να έχει σημαντικό κομμάτι της αγορά. Περισσότερο ποτέ τώρα η θάλασσα είναι προνομιούχος χώρος για τις βιολογικές παραγωγές. Δεν τυχαίο το ότι ο κανονισμός έφτασε ως κεραυνό εν εθρία τον Αύγουστο και χαιρετίστηκε θετικά. Αν και υπάρχουν πολλές αντιθέσεις εντός του κανονισμού, δεν θέλω να αντιπαράθεση στην την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται εμβάθυνση. Ο κανονισμό περιέχει τι διασυνδέσει, τη συμβίωση μεταξύ εγκατάσταση βιολογική και μη βιολογική. Και αυτό θα σημαίνει ότι σχεδόν τίποτα δεν κάναμε. Ο κανονισμό λοιπόν υπό το φω και των δικών μα σκέψεων μπορεί, μπορεί, μπορεί λέγω να προτείνει να προταθεί τροποποίηση αλλαγή του κανονισμού, τόσο ώστε να υπάρχουν αυστηρότερε προποθέσει και διατάξει όσον αφορά τι βιολογικέ υδατοκαλλιέργειε. Χρειάζεται και ένα σήμα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση Βιολογικό Προϊόν. Ένα σήμα που θα στηρίζεται μέσω των αυστηρών ε, επιλογών που προβλέπει ο κανονισμός όσον αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων και διαφόρων συνθήκων που προβλέπονται. μέσω ρυθμίσεων που προβλέπουν την καλύτερη υγεία των ίδιων των ηχθείων. Προβλέπουμε κάτι για την υγεία των πουλερικών και δεν ασχολούμαστε με την υγεία των ψαριών, εις κλοβούς. Ίσως δεν ακούμε με τα αυτιά μας τις κραυγές τους γι' αυτό. Αλλά και οι τεχνικές μεταφοράς των ψαριών και εισόδου των ψαριών στους κλοβούς εκεί των ηχθείων πρέπει να είναι κάτι που να προβλέπεται. Όπως και η χρήση ελεγχόμενη των φαρμάκων η περίπνηση και έλεγχος αυτών και πώς μεταφέρονται όλα αυτά μέσω της τροφικής αλυσίδας. Μόνο κόβοντας αυτούς τους γόρδιους δεσμούς και με αυστηρές προδιαγραφές και με το ευρωπαϊκό σήμα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη σωστή προσέγγιση για την αγορά. Ανταγωνιστικότητα. Να πουλείτε, να σαν καλό προϊόν στη διεθνή αγορά το προϊόν μας. και να, και να δημιουργηθεί ένα σημείο, να είναι σημείο ισχύος ο κανονισμό για την εισαγορά. Να είμαστε πιο αυστηροί στην νομοθεσία μα όσον αφορά τα, τα προϊόντα που εισάγονται ταυτόχρονα. Εξαιρετικά συνοπτικά τα παρουσίασα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ε, ίσως να μπερδεύτηκαν με αυτά που είπα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η περίοδος που έχουμε μπροστά μας, ε, το, χρόνο, χρόνος που έχουμε μπροστά μας θα μου δώσει τη δυνατότητα να δεχθώ συστάσεις σας και να ανταλλάξουμε απόψεις. Βάσει αυτού θα ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα εργασίας. Ακολουθήσει μια συζήτηση. Παρουσίαση των μελετών που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχέ Νοεμβρίου, 3 και 4 Νοεμβρίου θα γίνει αυτό. Θα υπάρξει και ένα έγγραφο εργασία που θα αποσταλεί στι μεταφραστικέ υπηρεσίες 13 Νοεμβρίου, παρουσίαση στην Επιτροπή, στην Επιτροπή, πρώτη παρουσίαση του εγγράφου στην Επιτροπή, θα λάβει χώρα στι 30 Νοεμβρίου. Μια μακρά φάση, μια παύση θα έλεγα, θα ακολουθήσει λόγω της επιλογής των επιτρόπων κλπ. Μετά θα γίνει ακρόαση στις 16 Μαρτίου και θα υποβραθεί η έκθεση στην Επιτροπή 7 και 8 Απριλίου για να υιοθετηθεί στην Επιτροπή 4 Μαΐου και να φτάσουμε στην Ολομέλεια στη Σύνοδο του Μαΐου. Αυτή είναι η διαδρομή. Αρκετά μακρά διαδρομή. Έτσι, αυτή η δουλειά που ξεκινά μόλις σήμερα και παρόλο που είναι η πρώτη φορά που εκλέγομαι βουλευτής και για πρώτη φορά μέλος της Επιτροπής αυτής, λέμε κάθε ταπεινότητα. Σας ζητώ λοιπόν να βοηθήσετε, ούτως ώστε η δουλειά μου να καταλήξει σε καλά αποτελέσματα. Δεν έχει μείνει και τόσο ε, χρόνο να αρχίσουμε αυτή την κουβέντα. Και κύριε Προσέδο, δεν έχουμε χρόνο, παρακαλώ. Σε ένα λεπτό και κατόπιν άλλο ένα λεπτό θα ε, λάβω εγώ το λόγο και άλλο ένα έχει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και θα είμαι τηλεγραφικός, μια που έχουμε τα θέματα τόσο σημαντικά και αντιφατικά μεταξύ τους. Υπάρχει εδώ πέρα πρόβλημα με την ηχθειοκαλλιέργεια. Αυξάνει η ζήτηση και έχει μέλλον ο κλάδο. Όμω θα πρέπει να υπάρχει μια ανάπτυξη που να γίνει βιώσιμα. Και γι' αυτό και συμφωνώ ότι χρειάζεται κάποιο πλαίσιο για την εξέλιξη αυτή, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Και να υπάρχουν επίση ε, νομοθετήματα, να υπάρχει μια στρατηγική, να αφορά την ε, ποιότητα, τόσο ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε την αυξανόμενη διεθνή ε, τάση ανταγωνισμού, να προστατεύσουμε, να δώσουμε ποιοτικό προϊόν στου καταναλωτέ να υπάρχει έρευνα, τόσο ώστε να μπορέσουμε να, να, να διαφοροποιηθούμε, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα και γι' αυτό και θα πρέπει ε, ξεκάθαρα να δούμε πού θα εγκαθίστανται οι σχετικοί, αυτοί που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, να υπάρχει αρμονία σε σχέση με το περιβάλλον μας και να μην ε, υπάρχει μονομερής ανάπτυξη, μην υπάρχει αυθαιρεσία, ε, να υπάρχει ευταξία και βέβαια αυτό να γίνει μέσω της επικουρικότητας με την καλή έννοια. Και είναι αυτό που λέμε προσθετικότητα. Και επίση θα πρέπει να τηρείται το κοινοτικό δίκαιο, σχετικέ διατάξει, οι εθνικέ διατάξει και ό,τι γενικά ε, είναι προ το συμφέρον των περιφερειών. Και έτσι θα έχουμε αρμονική ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη αυτού του κλάδου, χωρί να θέτουμε κινδύνο το περιβάλλον με κάποιε δραστηριότητε που είναι δυνατόν να καταλήξουν σε ε, κάποια ένταση για κάποιο χώρου, για κάποια περιβάλλοντα που κρίνονται άξια προστασία. Και βέβαια για να γίνει μια τέτοια στρατηγική ε, εφικτή θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι πόροι για να δώσουμε την κατάλληλη όθηση στη στρατηγική μας. Τώρα, θα ήθελα να σας πω πολλά, αλλά θα σας πω ένα πράγμα μόνο τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την συνεδρίαση. Αυτό που είπατε για τις δαπάνες, για την ε, ποιότητα, γιατί είναι κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό το οποίο υπάρχει σε αυτήν την εκθέση, ότι δηλαδή οι εισαγωγέ, πάρα πολύ σωστά είπατε, αυτέ που έχουμε από τι τρίτε χώρε ε, και για τα προϊόντα εκθεοκαλλιέργεια, μιλώ πολλέ φορέ, δεν συμμορφώνονται με κάποιε διατάξει που αφορούν στους δικούς μας παραγωγούς. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική προτίμηση, αλλά μπορούμε να υποχρεώσουμε τις τρίτες χώρες να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις που τάσουν και εμείς τους δικούς μας. Κυρία Συγγετρή, έχετε για ένα λεπτό το λόγο. Το ξανάχασα. Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις σας και τα σχόλιά σας. Φυσικά θέλετε συνεργασία. Εγώ απλώς θα ήθελα να δώσω κάποιες έτσι, γενικές αρχές Απ' την άλλη δεν έχουμε πολλά αλλιεύματα. Πάντα εισάγουμε. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Όχι μόνο για οικονομικούς λόγους βέβαια. Αλλά και για την... για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες προσφοράς και ζήτησης. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα, τα προβλήματα που υπάρχουν με την υδατοκαλλιέργεια, με, τους, ε, με όσους εμπλέκονται σε μίσο ποσο ο τουρισμός, ε, το περιβάλλον κλπ. Η offshore υδατοκαλλιέργεια είναι ένα τομέα που πρέπει να δούμε. Βέβαια, πολλέ φορέ ε, θεωρούμε ότι εντάξει, δεν είναι κανένα σημαντικό τομέα, δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον, ε, απασχολούνται εξειδικευμένοι άνθρωποι, υπάρχει καταλληλή κατάρτιση. Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αυτό είναι και πηγή ε, εισοδήματος για τους αλληλείς. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα προϊόντα, γιατί οι καταναλωτές δεν έχουν πάντα ειδική ε, έτσι, άποψη για τα προϊόντα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Κύριε Ευχαριστώ. Δύο γρήγορε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, το κεφάλαιο 5-9 τη Πράσινη Βίβλου για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική θέτει το ζήτημα του ρόλου τη υδατοκαλλιέργεια στη μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική. Αυτό το θέμα είναι κατά πώ θα πρέπει να ενταχθεί αυτή η δραστηριότητα στην κοινή αλληλευτική πολιτική με συγκεκριμένους στόχους και ειδικά εργαλεία που αυτή ήταν η επιλογή παρουσίασε ο εισηγητή που πιστεύει ότι πρέπει να γίνει γενικό το, τομεακό κανονισμό που θα συμπεριλαμβάνει όλε τι πτυχέ δραστηριότητα. Μία λύση αυτή. Άλλη επιλογή. Τα κράτη-μέλη να φροντίσουν επιθνική σε εθνικό επίπεδο να βρουν τη λύση. Αυτή είναι η παρούσα κατάσταση. Από εκεί έχει ελάχιστε αρμοδιότητε η κοινότητα όσον αφορά τι εθνοκαλλιέργειε. Είναι στο επίκεντρο το θέμα αυτό τη κοινή αλληλευτική Πολιτική και ο συγητής εξέφρασε κάποια προσέγγιση και περιμένουμε την έκθεση τη επιτροπή αυτή και του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η θέση σας όσον αφορά αυτά τα θέματα. Δεύτερη παρατήρηση. Εντοπίσαμε το βασικό πλαίσιο των περιορισμών τη ετοκαλλιέργειας, που είναι η έλλειψη χώρου ανάπτυξη. Δεν δίνουν πλέον άδειε για ετοκαλλιέργεια τα κράτη-μέλη. Μπορούμε να μιλάμε για έλλειμμα όσον αφορά τα ψάρια στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ανάπτυξη το για καλλιέργειο. τα κράτη-μέλη δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι γεγονό. Είναι μεγάλο ε, περιορισμό για την ετοκαλλιέργεια και από τη στιγμή που δεν αλλάζει αυτό και έχετε πραγματική εξουσία να επηρεάσετε εσεί την κατάσταση, η ετοκαλλιέργεια δεν θα αναπτυχθεί σύμφωνα με την ανάλυση μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία κύριε μάλλον, δεν έχουμε χρόνο θα πρέπει να αρχίσουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Όσοι θέλει το λόγο, παρακαλώ να μιλήσει ε, στην επόμενη συνάντηση, στις επόμενες. Κύριε εισηγητή. Και εγώ θέλω ένα λεπτάκι. Οι παρατηρήσεις όλες ήταν ακριβείς. Δύο ερωτήσεις, δύο θέματα. Πράγματι, η κοινότητα δεν έδωσε επιλογές στα κράτη και δεν είναι όριμο ο κανονισμό σήμερα. Γιατί να κάνουμε έναν κανονισμό, λοιπόν, ερωτώ για την υδατοκαλλιέργεια τη βιολογική. Υπάρχει αντίφαση. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Πιστεύω ότι οι παρατηρήσει όλε ήταν επίκαιρε. Εγώ συνοπτικά λέω ότι συμμερίζομαι αυτά που υπόθηκαν. όσον αφορά το σεβασμό της ποιότητας, το σεβασμό της πρόσβασης των, ε, στα προϊόντα στην Ευρώπη. Είχα να πω πολλά, αλλά συνοπτικά τα παρουσίασα. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειε. Τα διοικητικά θέματα θα πρέπει να βρουν λύση. Εξού και η, ανάγκη που υπάρχει. Πιστεύω ότι να αφήσουμε στα κάτι μελη το θέμα της διοργάνωσης αγοράς οδήγησε σε περιορισμούς και όρια όσον αφορά τις περιβαλλοντικές συνέπειες και μη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα της κοινή ε, δράσης. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά αυτά. Δεν έχουμε χρόνο, κλείνω εδώ και όποιο έχει παρατηρήσεις δεν είναι γενική πρόσκληση. Ουσιαστική πρόσκληση είναι επειδή συζητήσαμε ελάχιστα, παρακαλώ να μου στείλετε κάποιες προτάσεις κλπ. για να το ανταλλάξουμε απόψεις. Lana, y pido disculpas de verdad, pero a las cinco y media teníamos... Συγγνώμη, συγγνώμη πραγματικά, πεντέμιση πρέπει να έχουμε αρχίσει την ένδυση των συντονιστών. Συγγνώμη από δεν μπορούσαν να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ, ε, αποχωρήσατε οι υπόλοιποι.